So, ε, συνάδελφοι, αρχίζουμε λέει ο πρόεδρος. Ε, ως συνήθως από το υπαρθμό ένα αρχίζουμε που είναι η έγκριση μερικές διατάξεως και σας προτείνω τα σημεία 3 και 16 να αναβληθούν. Uh, το 10 δε είναι μια ψηφοφορία. Αφορά την 30η Μαΐου, αλλά αναβάλλεται, όμως θα συνεχίσει να ισχύει η προβληπόμενη συζήτηση για τις 29 Μαΐου, σήμερα δηλαδή. Τώρα η παρουσίαση των ε, καθεντήριων γραμμών όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 141 του καταστατικού ε, αναβάλλεται, ήταν ε, ε, και κλεισμένο να συζητηθεί. Επίσης, ο κύριος Καβαντά, το 9, μια ψηφοφορία και το έτοιμο του κύριου Καβαντά εγκρίνεται και θα αναβληθεί αυτή η ψηφοφορία. Έχει κάνει ένσταση για αυτές τις αλλαγέ. δεν βλέπω κάποιον να ενίσταται. Μετά, δύο, ανακοινώσει του Προέδρου. Δεν έχω τίποτα να σα ανακοινώσω και συνεχίζουμε. Έχουμε το θέμα υπαριθμών 4. Συζήτηση του σχεδίου έκθεσης όσον αφορά τους κανόνες για άσκηση δικαιωμάτων δημιουργού συγγενικών δικαιωμάτων. Επίσης και τον λόγο έχει ο κύριος Βόλκεν που είναι ο συγγητή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα γερμανικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά την ε, έκθεση αυτή, πρόκειται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ε, σε τηλεοπτικούς σταθμούς και φυσικά την ολοκλήρωση και την ε, η ύπαρξη μιας πραγματικής ψηφιακής αγοράς, να μην υπάρχουν πλέον εμπόδια και σύνορα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να μπορεί να υπάρχει μεταφορά δεδομένων ψηφιακών με έναν απρόσκοπτο και εύκολο τρόπο. Να μην υπάρχουν εμπόδια και αν αυτό επιτευχθεί, Φυσικά προϋπόθεση είναι να υπάρχει η νομοθετική, νομική λύση όσον αφορά τον κανονισμό, τον οποίο όπως ξέρετε έχουμε συνηθίσει. Γιατί αναφέρθηκα καταρχήν στον κατακαιρματισμό το νομικό και γιατί αναφέρθηκα επίσης και σε αυτό το οποίο ονομάζουμε κατακαιρματισμό της ψηφιακής αγοράς. Η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά όσον αφορά τις διασυνοριακές μεταφορές δεν μπορεί να υπάρξει διότι όπως ξέρετε υπάρχει μία, ένας, ε, ένα είδος εμποδίων στα σύνορα τα προγράμματα παραδείγματο χάρη του ενός ραδιοφωνικού σταθμού όσο κοντά να βρίσκεται στα σύνορα μιας άλλης χώρας δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά οι πολίτες των γειτονικών χωρών. Πολλά προγράμματα μεταφέρονται και μεταδίδονται μόνο με το διαδίκτυο, δεν μπορούν δηλαδή να μεταδοθούν με τον ε, παραδοσιακό τρόπο, υπάρχει δηλαδή μόνο η γραμμική μετάδοσή τους, κάτι που δεν επιτρέπει την παραδοσιακή τους μετάδοση παρά μόνο με ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δυστυχώς οι εθνικές άδειες είναι κάτι που παραμένουν δεν έχει ακόμα γίνει αποδεκτή η ιδέα των διεθνών αδειών και θα ήθελα να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Θα αναφερθώ ιδιαίτερα στο άρθρο 1, Β της ε, οδηγίας για τους δορυφόρους, κάτι που αναφέρει πολύ συγκεκριμένα στην αρχή της χώρας προέλευσης. Και βεβαίως εγώ γνωρίζω ότι είναι πολύ σημαντικό εδώ να υπάρχει ε, το θέμα των κινηματογραφικών ε, παραγωγών, κάτι που θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσει να υπάρχει η ο πλούτος της ε, καλλιτεχνικής δημιουργίας και να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην Ευρώπη ε, σε αυτά τα ε, καλλιτεχνικά δημιουργήματα, στα έργα τέχνης, του κινηματογράφου. Και ακριβώς αυτό προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε με αυτόν τον κανονισμό. Να υπάρχει δηλαδή ποιοτική και ποσοτική ελευθερία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει αυτή η ενιαία αγορά, κάτι που θα δώσει νέες δυνατότητες ανάπτυξης τη δημιουργικότητα στην Ευρώπη. Θέλουμε πραγματικά και πρόκειται για μια καθαρά πολιτική ε, ε, έκθεση να δείξουμε ότι όλα αυτά τα τεχνικά θέματα δεν ε, είναι απλή τεχνολογία αλλά πίσω από αυτές τις προσπάθειες υπάρχουν δημιουργοί, υπάρχουν άνθρωποι ε, που θέλουν να προωθήσουν μηνύματα, έργα τέχνης, άνθρωποι που ζουν κοντά στα σύνορα και οι οποίοι θέλουν ελεύθερη πρόσβαση σε καλλιτεχνικά ε, περιεχόμενα και δεδομένα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Η πρόσβαση σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό μιας άλλης χώρα είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Είναι λοιπόν σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι το 35% είναι ακριβώς αυτό που προτείνουμε εδώ για το περιεχόμενο τις κοινοπραξίες αυτές για την μειοψηφία των μετόχων. Θέλουμε κάθε φορά να εκπροσωπούμε τους καταναλωτές, τους Ευρωπαίους πολίτες και όπως ακούσαμε και κάθε φορά που συζητήσαμε με τις ομάδες συμφερόντων, αυτές οι ιδέες θα πρέπει να προωθηθούν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς βεβαίως θέλουμε να ακουστούν όλες οι νέες ιδέες για την μεταφορά δεδομένων, και θα ήθελα να αναφέρω επίσης και θέματα ανταγωνιστικότητας. Το δίκαιο του ανταγωνισμού, παραδείγματο χάρη, είναι κάτι το οποίο αναφερθήκαμε πολλές φορές. Εδώ βεβαίως υπάρχουν περιορισμοί σε κάποιο είδους ελευθερίες όταν ε, παραβιάζονται οι κανόνες του ανταγωνισμού. Αλλά βεβαίως τα πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να να προστατεύουν, συγγνώμη, εδώ αποκλειστικά και μόνο τον δημιουργό, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά και οι αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και σε κάθε κράτος μέλος όταν υπάρχουν διαφορετικοί ε, ραδιοφωνική σταθμή, τηλεοπτικά κανάλια τα οποία εκπέμπουν σε γειτονικές περιοχές, σε ε, άλλα κράτη-μέλη, να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, να ισχύει η ίδια νομοθεσία. Βεβαίως, ξεχνάμε πολλές φορές ότι υπάρχουν και κάποια άλλα συμφέροντα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε περιπτώσεις ε, συγχωνεύσεων, παραδείγματος χάρη, και το θέμα των εμποδίων που χρησιμοποιούνται σήμερα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα κανάλια της τηλεόρασης δεν θα πρέπει να λειτουργούν παραβιάζοντας τις αρχές του ανταγωνισμού. Χρειάζεται νόμιμη πρόσβαση, νόμιμη πρόσβαση στα περιεχόμενα αυτών των αυτό ήταν εξάλλου και το νόημα των τροπολογιών που έχω υποβάλει. Τι μας ενδιαφέρει, να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή παραγωγή. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κύριο μέλημά μας. Εγώ θέλω να στηρίξω την ευρωπαϊκή παραγωγή και νομίζω ότι αυτό, αν διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο που σας παρουσιάζω, θα το αντιληφθείτε. Και αυτό φαίνεται εξάλλου και στο άρθρο 2.2 η τροπολογία 15, η τροπολογία 19, καθώς και άλλες τροπολογίες που ζητούν νέες αποδοχές. Είναι κάτι που στον κινηματογραφικό τομέα, παραδείγματο χάρη, θέλουμε να προστατευθεί η ε, κατηγορία των δημιουργών, των ηθοποιών, καθώς και ένας δίκαιος τρόπος αμοιβή τους. Βεβαίως σήμερα θα πρέπει να κοιτάξουμε και τις προοπτικές ε, του μέλλοντος. Βεβαίως η τεχνολογία εξελίσσεται και θα πρέπει να υπάρξει μια νομική ασφάλεια η οποία να εγγυάται τις ε, μελλοντικές αυτές τεχνολογικές εξελίξεις και πώς θα προβλέψουμε την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα αυτά, καθώς και κάποια άλλα περιεχόμενα τα οποία μπορεί κανείς να τα βρει μόνο online. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ε, κάποιες συγκεκριμένοι περιορισμοί στις ελευθερίες και αυτό νομίζω ότι μετά από τη συζήτηση που ακολούθησε στην τελευταία μας παρουσίαση μπορεί να οδηγήσει σε κάποια αποδεκτά από όλους ε, ε, πακέτα προτάσεων και για τις αμοιβέ, αλλά και για την τροπολογία 17 και την χώρα προέλευσης. Εγώ ήθελα πραγματικά να αποφύγω το να στηρίξουμε κάποιες χώρες περισσότερο. Γι' αυτό και η τροπολογία 17 έχει ακριβώς αυτό το περιεχόμενο. Να μην υπάρχουν καταχρήσεις από κανέναν. Πολύ σημαντικό είναι επίσης ε, το θέμα του περιεχομένου, όπως σας είπα, είτε αυτό βρίσκεται online είτε όχι, αλλά και η μετάδοση καλωδιακή στην τροπολογία 21 και στις επόμενες βλέπετε τις προτάσεις αυτές που αφορούν την καλωδιακή μετάδοση. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά τον ε, κανονισμό αυτό που αφορά και την φορητή μετάδοση είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το αναπτύξουμε ιδιαίτερα. Επιμένω σε κάθε περίπτωση στο ποσοστό του 30%. Επιμένω ότι το περιεχόμενο και η ευρωπαϊκή συνιστόσα θα πρέπει να προστατευτεί. Ολοκλήρωσα με τις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, ε, Ευχαριστούμε πολύ, η κυρία Ρέντα. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή, γιατί μας εξήγησε πόσο σημαντική είναι αυτή η πρόταση για τους καταναλωτές. Είναι σαφές ότι κάτι θα πρέπει να γίνει. Να νομοθετήσουμε ούτω ώστε αυτόν τον υγειοαποκλεισμό να τον αντιμετωπίσουμε γιατί αυτή η γεωγραφική φραγή τώρα εμποδίζει τους καταναλωτές και πάρα πολλές φορές οι καταναλωτές αν δεν θέλουν να πληρώσουν για πρόσβαση σε κάποιο περιεχόμενο, ε, τότε δεν μπορούν νόμιμα να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό με οποιαδήποτε μορφή. Α δούμε ποια είναι η αντίδραση των εμπλεκομένων. Ε, από αυτήν φαίνεται το πόσο σημαντικό είναι το θέμα και είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλουν οι φορείς, υπάρχει να το εντοπίσουν. Τόσα χρόνια έχουμε προσπαθήσει με διάφορα νομοθετήματα και δεν βελτιώθηκε ουσιαστικά η κατάσταση. Επομένως ήρθε η ώρα κάτι να κάνουμε νομοθετικά και αυτό είναι το τμήμα της δέσμης των μέτρων Έτιγκερ του φθινοπόρου. θα πρέπει να μην σχετίζεται με συγκεκριμένη επικράτεια, το copyright κλπ. Όσον αφορά το σχέδιο της έκθεσης, είναι μια σωστή βάση αφετηρίας ε, συζήτησης. Έχουμε κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα-πρώτα για τον ορισμό των Ιντερνετικών υπηρεσιών θα πρέπει εδώ να καλύψουμε και κάποιο υλικό το οποίο διατίθεται πριν ή μετά την εκπομπή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ε, προγραμμάτων για να καλύψουμε και κάποια τα προγράμματα τα οποία έχουν φτιαχτεί για το ίντερνετ. Και αυτό προς το παρόν δεν καθίσταται σαφές από τον ορισμό του εισηγητή. Λέει για περιεχόμενο το οποίο εμπλουτίζει ή διευρύνει την εκπομπή, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά ευρύ, γιατί μπορεί να υπάρχουν ε, κάποιο είδους έργα, τα οποία φτιάχτηκαν για το ίντερνετ και να μην σχετίζονται άμεσα με κάποιο είδου εκπομπή και μετάδοση εκτός ίντερνετ. Άρα κάτι να κάνουμε τον ορισμό για να καλύψουμε και αυτά. Ο σχέση και να υπάρχει με ε, εκπομπή περιεχομένου εκτός. Τώρα για την αναμετάδοση, θερμεδοουδέτερη ε, μετάδοση και να καλύψουμε τις αναμεταδόσεις ε, με το ίντερνετ, με τη διεύθυνση IP. Και έχουμε τώρα και κάποιε άλλες προβληματικές διατάξεις στα όσα προτείνει παραπέρα ο Εκεί που λέει ότι δεν μπορεί κανεί να απεμπολίσει τα δικαιώματα σε αμοιβή. Καταλαβαίνω την καλή του πρόθεση να εξασφαλίσει δηλαδή ότι πάντοτε θα καταβάλλεται ένα αντίτιμο εάν ε, κάποιος πάρογος όμως διέπεται μια τέτοια διάταξη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί ε, ιντερνετικά να εκπέμψει κάποια ε, προγράμματα επί των οποίων έχει απεμποληθεί το δικαίωμα σε αμοιβή. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρη κατά πόσον αυτό είναι ο κατάλληλος τρόπος να λυθεί το πρόβλημα γιατί υπάρχουν και κάποιες διατάξεις όσον αφορά την έγκριση κάποιων μεταδόσεων που είναι διασυνοριακές και αφορούν την ε, αμοιβή. Επίσης, άλλη μια επίκριση ότι στο σχέδιο κειμένου έχουμε πολλές εξαιρέσεις για την αρχή της χώρας προέλευσης. Πρώτα-πρώτα η εξαίρεση που αφορά τους παρόχους περιεχομένου που στοχεύουν βασικά σε κάποιες χώρες εκτός των χρόνων μελών τους. Εκτός των χρόνων μάλλον που είναι εγκατεστημένοι υπάρχει. Και οπότε θα πρέπει να δούμε το πώς κανείς δεν θα ψάχνει το πιο ευνοϊκό καθεστώς σε άλλη χώρα και να δούμε κατά πόσον κάποιο ε, πάροχος μετεγκαθίσταται και πάει σε άλλη χώρα μόνο και μόνο γιατί εκεί υπάρχουν πιο ευεργετικές ε, διατάξει για να κάνει τη δουλειά του. Νομίζω ότι περισσότεροι πάροχοι έχουν τη βασική τους λειτουργία και τα βασικά τους εισοδήματα τα έχουν εκτό ίντερνετ. Άρα μήπω και δεν χρειάζεται αυτή η διάταξη. Μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτή η εξαίρεση για την πιο μακρά περίοδο ισχύω για τα κάποια έργα, κάποια κινηματογραφικά έργα. Εδώ ποιος είναι ο κίνδυνος. Η Ιντερνετική πάροχη, ιδίως για τους πιο νέους χρήστες, δεν μπορούν τίποτα να κάνουν γιατί αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν κάποιες πλατφόρμες on demand. Και αυτές οι υπηρεσίες δεν τις δικούν στα όσα θέλουν οι χρήστες. Αυτές οι πλατφόρμες VOD όπως το Netflix. Πριν από τρία χρόνια τίποτα δεν υπήρχε από αυτά. Είδατε επομένω πόσο γρήγορα εξελίχθηκαν τα πράγματα σε μία τριετία. Άρα αυτή η θέση σε ισχύ να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα η ιδάλλως. Θα είναι απαρχιωμένος ο κανονισμός και πριν ακόμα τεθεί σε ισχύ και θα θέλει επικαιροποίηση. Άρα, όλα αυτά θα συζητήσουμε τον εισηγητή, ελπίζουμε όλα πάνε καλά και θα κατεβάσουμε και κάποιε τροπολογίε για να διορθώσουμε τα σημεία που σα εξηγήσαμε. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το κείμενο αυτό, για την εργασία του επιτυχημένου αυτή που είναι περίπλοκο ε, και δύσκολο. Ε, είχα και εγώ αυτή την εμπειρία γιατί το συζητήσαμε και στην Επιτροπή ε, ΙΜΚΟ. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για πολλά καλά πράγματα, όπως για παράδειγμα την επέκταση της συλλογικής διαχείρισης για τις over-the-top υπηρεσίες για τους φορείς καλωδιακής τηλεόρασης ώστε να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση βάσει του είδους της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Αυτό είναι μια προσαρμογή την οποία επικροτούμε ε, και κάτι ακόμη που είναι αρκετά τεχνικό επίση, ότι έχει να κάνει με την άμεση έγχυση, δηλαδή πώς μπορούμε δηλαδή να ε, υπάρχει ένα πρώτο πρόγραμμα ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και στη συνέχεια μια αναμετάδοση, το ίδιο ε, το δικαστήριο δεν ξέρει ακριβώς την επιχειρησιακή πραγματικότητα πώς να την μεταχειριστεί, άρα είναι χρήσιμο αυτό που προτείνει ο εισηγητής και τον ευχαριστώ πολύ. Βέβαια υπάρχει το βασικό ε, ζήτημα της αρχής ε, χώρας προέλευσης που δημιουργεί ε, προβλήματα βεβαίως πολύ σοβαρότερα πολύ σημαντικότερα από τις τεχνικές αυτές προσαρμογές. Πρέπει κάποια στιγμή να αναρωτηθούμε πώς ε, λειτουργεί ολόκληρος ο ραδιοτηλεοπτικός, ε, οπτικοακουστικός τομέας, ε, οι σκηνοθέτες, η παραγωγή ταινιών, όλοι οι φορείς μετάδοσης. Μιλάμε δηλαδή για τη μετάδοση κάποιων ε, έργων στο διαδίκτυο, όμως το πρόβλημα που υπάρχει είναι η εδαφική ε, αποκλειστικότητα. Μπορεί να ε, θεωρούμε ότι είναι ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο κάποια στιγμή θα εξελιχθεί στο μέλλον, αλλά σήμερα για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την οπτικογραφική παραγωγή πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα σε όσους κάνουν την παραγωγή να έχουν κάποια επιστροφή στην επένδυσή τους και αυτό το κάνουμε μέσω του εδαφικού αποκλεισμού το να μπορέσουμε λοιπόν ε, να ε, δώσουμε, να δοθούν κάποια δικαιώματα ε, βάσει πολύ συγκεκριμένων αρχών, ανάλογα με τη χρονική στιγμή, ανάλογα με το πού που γίνεται η αναμετάδοση, είναι μία πραγματική αποδυνάμωση όλων όσων είναι δημιουργοί των οπτικοακουστικών αυτών έργων ε, υπέρ όλων αυτών που είναι υπεύθυνοι μετάδοση και στη συνέχεια αναμετάδοση. Οπότε λοιπόν εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τον οπτικοακουστικό τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όμω αυτή η αποδυνάμωση ε, τη ε, συμβατική σχέση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων είναι ε, κάτι το οποίο τελικά ε, δεν βοηθά ούτε τους δημιουργούς, ε, γιατί θα καταλήξει σε ακόμη περισσότερη μείωση ε, των εσόδων τους. Ε, ενδεχομένως ε, να θέλουμε να υποστηρίξουμε κάποιους των οποίων η οικονομική αποδοτικότητα δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά πάρα πολύ σημαντική από απόψεως ευρωπαϊκών αξιών και οι πιο μικροί ακριβώς που εξασφαλίζουν την ευρωπαϊκή ποικιλομορφία είναι αυτοί οι οποίοι θα αποδυναμωθούν, θα βρεθούν σε μια μειονεκτική θέση βάσει αυτής της αρχής της χώρας προέλευσης. Πραγματικά ε, αποδυναμώνει μου τη θέση τους ε, και πραγματικά πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά ακόμη για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη δουλειά που πρέπει να γίνει. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες του εισηγητή. Θεωρώ ότι το κείμενο είναι μια καλή βάση. Σωστά πρέπει να προβληματιστούμε για μερικά σημεία παραπάνω. Ε, Κύριε Καβαντά, να σας συγχαρώ για ε, όσα είπατε για τον κανονισμό περί της, ε, ε, του, να μπορούν να μεταφερθούν τα δικαιώματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από μερικές εβδομάδες ψηφοφορία στην Ολομέλεια δεν έχει νόημα να εξετάζουμε ένα κείμενο το οποίο θα θέσει να αμφιβόλο όλα αυτά τα οποία καταφέραμε μέσω της έκθεσής σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ για την κυρία Λεκρίπ, <clears throat> θα ήθελα να πάρω το λόγο καταρχήν. Είναι σκιώδης η συγγήτρια. Θα πω λοιπόν στα αγγλικά αυτά τα οποία μου έδωσε. Θέλω να μας πεντιμήσει αυτά που ήδη είχε εκφράσει σχέση με τον κανονισμό, το θέμα της αφαιρότητας ε, της ε, δημιουργικότητας στην Ευρώπη, υπονομεύοντας το θέμα των αδειών και της εδαφικής στήριξης αυτών των αδειών. Όσον αφορά τώρα την συγκεκριμένη έκθεση, η κυρία Λεγκρίφ πιστεύει ότι το θέμα της αμοιβή που βασίζεται, για τους δημιουργούς που βασίζεται ε, στο κράτος προέλευσης δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβαδίζει με, την ε, παρούσα, με τον παρόντα κανονισμό. Η κυρία Λεγκρίφ θέλει βεβαίως να συζητήσει το θέμα αυτό, είναι ανοιχτή συζήτηση, θεωρεί όμως ότι το άρθρο 2 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί, αλλιώ δεν θα μπορέσει η ομάδα του ΕΛΚ να στηρίξει το τελικό κείμενο. Όσον αφορά για το άρθρο 3, η πρόταση του εισηγητή είναι υπό εξέταση. Θεωρούμε ότι οι τροπολογίες εδώ είναι σωστές και θα συνεχίσω γιατί θα ήθελα να εκφράσω και τη δική μου άποψη και να προσθέσω κάτι. Αναφερθήκατε στο ερώτημα για ποιον κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν το κάνουμε μόνο για τους δημιουργούς, δεν το κάνουμε μόνο για τους καταναλωτές, για τους χρήστες. Το κάνουμε γιατί υπάρχει η στρατηγική της δημιουργίας μιας ε, ενιαίας αγοράς, ε, ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Βεβαίως και λαμβάνουμε υπόψη μας την στήριξη των δημιουργών, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά, αν θέλετε, και εξίσου σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη σε αυτό το κανονισμό. Όλα αυτά ε, με ισορροπημένο τρόπο. Γι' αυτό και θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι και για την παραγωγική και δημιουργική Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε στα πλαίσια αυτού του κανονισμού. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ όλων αυτών των πολλές φορές αντικρώμενων συμφερόντων κατά την άποψή μου και σε αυτό το τομέα θα πρέπει να τεθούν κάπως κάποια πολιτιστικά σύνορα. Υπάρχει ο Νότος, υπάρχει ο Βορράς με διαφορετικές πρακτικές, με διαφορετικές παραδόσεις. Πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας και γι' αυτό και μίλησα και για πολιτιστικά σύνορα. Από την άλλη, πιστεύω ότι βεβαίως και πρέπει να υπάρξει ελευθερία σύναψης συμφωνιών, αλλά αυτή η ελευθερία πρέπει να επεκταθεί και στις άδειες, και στην διάθεση στην αγορά. Και θα πρέπει βέβαια με τα νομοθετικά μας κείμενα να κατευθύνουμε αυτή την ελευθερία. Όσον αφορά τον οπτικό-ακουστικό τομέα, θα πρέπει να δούμε τι κινδυνεύει να προκύψει με αυτούς οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι και να στηρίξουμε αυτές τις κατηγορίες. Βεβαίως, η παραγωγή των ε, κινηματογραφικών έργων, οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, η στήριξή τους, η χρηματοδότησή τους είναι πολύ πιο εύκολη από μικρότερες παραγωγές. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε όλοι αυτοί οι οποίοι επενδύουν στις υποδομές, είτε επενδύουν στα περιεχόμενα αυτών των οπτικοακουστικών έργων, να γνωρίζουν με σαφήνεια τους κανόνες, πώς δηλαδή μπορούν ε, οι επενδύσεις τους αυτές, βάσει ποιων κανόνων, να έχουν ε, κάποιες ε, αποδόσεις. Γι' αυτό και πιστεύω ότι και το θέμα των τιμών, της απόδοσης μιας επένδυσης θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα παρουσιασμένο. Στην ε, πρόταση της Επιτροπής βλέπω ότι υπάρχει πρόταση για περιορισμό κάποιων δικτύων ε, και φορητών ε, αναμεταδόσεων, αλλά και βεβαίως αυτός ο περιορισμός των αριθμών των δικτύων μπορεί να έχει τελικά σαν σκοπό την ενδυνάμωση κάποιων δικτύων. Θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όπως είπα και προηγουμένως, με αυτούς που έχουν επενδύσει σε αυτές τις υποδομές και οι οποίοι θέλουν να γνωρίζουν το μέλλον ε, γιατί σαφώς και κάποια στιγμή θα χρειαστεί αναχρηματοδότηση, νέα χρηματοδότηση. Και βεβαίως μιλάμε για σχέδια πολιτιστικά. Όλα αυτά όμως από κάποιον χρηματοδοτούνται. Και αυτός ο οποίος επενδύει στον τομέα αυτό θέλει, επαναλαμβάνω, να γνωρίζει τους κανόνες. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν. Το διαδίκτυο, τα νέα κανάλια πρόσβασης, βεβαίως οι νέες τεχνολογίες Υπάρχουν κάποιες ρήτρε αποκλειστικότητας βεβαίως. Πρέπει να δούμε ποιες ε, τέτοιες ρήτρε θα παραμείνουν. Και επαναλαμβάνω, καλύτερη ισορροπία. Και σε καμία περίπτωση να μην κινδυνεύσουν κάποιες από τις δομές ε, οι οποίες θέλουμε να στηριχτούν. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να σας ζητήσω να είστε λίγο πιο σύντομοι γιατί δυστυχώς ε, δεν... Ε, έχουμε αρχίσει να καθυστερούμε επικίνδυνοι κύριε Καρύμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, πραγματικά έχω πολλούς ενδιασμούς σε σχέση με την ανάγκη ύπαρξης αυτής της πρότασης. Έχω ανησυχίε σε σχέση με ε, τη χρονική στιγμή της της πρότασης αυτής, ε, γιατί δεν έχουμε ακόμη δει ε, ποιος είναι ο αντίκτυπος σε σχέση με ε, το μοντέλο συγχρηματοδότηση και την απασχολησιμότητα στον τομέα αυτό. Επίσης, μόλις εγκρίναμε τον, τον κανονισμό για τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων εγώ πραγματικά έχω πολλού ενδιασμού σε σχέση με την έκκληση του για την επέκταση της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αρκετά μεγάλο βαθμό για να καλυφθεί και το ανοιχτό διαδίκτυο. Είναι σημαντικό για τους κάτοχους δικαιωμάτων να μπορούν να διαπραγματεύονται άδειε ε, μεμονωμένα, συμπεριλαμβανομένε επιπλέον αμοιβή μόνο για διαδικτυακέ υπηρεσίε. Νομίζω ότι θα αποδυνάμωνε την διαπραγματευτική ε, δυνατότητα των κατόχων δικαιωμάτων ε, θα έπρεπε να μην συμπεριλαμβάνεται ε, επιπλέον αμοιβή νομίζω λοιπόν ότι δεν υπάρχει λόγος να επεκταθεί η αρχή της χώρας προέλευσης στις διαδικτυακές υπηρεσίες ενδεχομένως μόνο στις ειδήσει η σωστή ισορροπία πρέπει να εξευρεθεί και ήδη πολλοί συνάδελφοι το ανέφεραν αυτό, η ισορροπία μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων και των καταναλωτών. Εγώ πραγματικά δεν έχω πιστεί ότι έχουμε πλησιάσει αυτό το στόχο σε αυτό το στάδιο. Ε, συνεπώς ε, θα υποβάλω τροπολογίες για να περιοριστεί ε, το πεδίο εφαρμογής ε, σύμφωνα με τα σχόλια που μόλις ε, σας έκανα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ο κύριος Καβαντά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, πάρα πολύ τον κύριο Φέλκεν ε, για το σχέδιο έκθεσης ε, που περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία αλλά και κάποια στοιχεία ανησυχητικά, ειδικότερα η θέση του σε κάποια θέματα τα οποία θα αναφέρω. Κάτραχας, το να εξετάσουμε το πρόβλημα της άμεσης έγχυσης περιεχομένου στην περίπτωση που ο φορέας ραδιοφωνικής μετάφωσης της κάνει μια έγχυση σε ένα κλειστό κύκλωμα. Ε, στη συνέχεια ο φορέας ε, το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό και μιλάω για την τροπολογία 8. Είναι κάτι που μου φαίνεται θετικό και λογικό. Όμως ε, είναι πολύ σημαντικό αυτά τα δύο μέρη να ε, είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενό τους και κάθε ένα από τα δύο μέρη να έχει ε, αδειοδοτήσεις και κάποια δικαιώματα για τους λόγους στους οποίους πολύ σωστά εξήγησε και η κυρία Ροζιέρ. Είναι πάρα πολύ απλός ο λόγος. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν κλάδο ψηφιακό και μια ψηφιακή αγορά πρέπει να υπάρχει κάτι το στέρεο στο εσωτερικό και αν ε, επηρεάσουμε την οικονομία αυτής της αγοράς, ε, ε, τότε είναι σαν να είμαστε συνένοχοι του ανοίγματο της αγοράς στην αμερικανική παραγωγή, ίσω και στην κινέζικη παραγωγή κάποια στιγμή. Ο Χρυσός Φίνικας δεν ήταν αμερικάνικος, ούτε σουηδικός, ούτε ε, κινέζικους και βέβαια είναι κάτι ε, το ε, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει κάπως να προστατεύονται. Μου φαίνεται ότι το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στόχο είχε σε μεγάλο βαθμό κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες, να δώσουν δηλαδή τη δυνατότητα κάλυψης κάποιων υπηρεσιών στο διαδίκτυο, πολύ συγκεκριμένων, όμως ο κύριος Βόλκεν θέλει να το διευρύνει αυτό για να συμπεριληφθεί ένα φάσμα πολύ ευρύτερο προϊόντων ε, στο διαδίκτυο και πρόκειται για την τροπολογία σας 12. Συμφωνώ και στο βαθμό στον οποίο αυτές οι υπηρεσίες... Ε, ε, είναι συγκρίσιμες ε, με κλειστού κυκλώματος υπηρεσίες, ε, τις υπηρεσίες για παράδειγμα όπως οι υπηρεσίες τηλεόρασης μέσω ίντερνετ. Όσον αφορά τώρα την αρχή της χώρας προέλευσης, εγώ συμφωνώ με κάποιους από τους προλαλήσαντες, είμαι εντελώ αντίθετος, κάτι το οποίο είναι περίεργο γιατί είναι ένα γερμανικό προνόμιο το οποίο δύο Γερμανοί ε, εισηγητές από δύο διαφορετικές ε, ομάδες προσπάθησαν να προωθήσουν ε, πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση γιατί εγώ είμαι παραδοσιακά φίλος και δεν έχω κανένα πρόβλημα συνήθως. Τώρα λοιπόν θα αντιταχθώ. Δεν βλέπω λοιπόν για ποιο λόγο θα έπρεπε να επηρεάσουμε τα πράγματα υπέρ ενός γερμανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα ε, δημόσιου. Ε, όσον αφορά την ε, αναζήτηση της καλύτερης, του καλύτερου καθεστώτος, του ευνοϊκότερου καθεστώτος, θα έπρεπε να ε, μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σοβαρές δικλείδες ασφαλείας. Εγώ δεν αρνούμε αυτό το οποίο ε, προτείνεται ε, κύριε Σιγητά, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποια ασφάλεια, κάποια δικλείδα ασφαλείας για να μην ξεφύγουν τα πράγματα. Όσον αφορά την αναμετάδοση τώρα, η αναμετάδοση είναι ένα ζήτημα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης ε, προσοχής και επιφυλάξεων ε, γιατί έχει να κάνει με το άρθρο 22 και το κείμενο 133 άρθρο 16 που δημιουργεί πρόβλημα ε, και που ζητά συμμετοχή του συνομοθέτη. Καταλαβαίνω ότι δεν έχετε αρκετή απόσταση για να μπορείτε να καταλάβετε ε, περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Ε, όμως εγώ ε, θα προχωρήσω σε τροπολογίες που θα έχουν σκοπό να αποκαταστήσουν αυτά τα οποία είπε το δικαστήριο και τα οποία θεωρώ ότι είναι καλύτερα για τον οπτικοακουστικό κλάδο της Ένωσης. Όσον αφορά την επιπλέον αμοιβή για τους δημιουργούς, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο. Καλό είναι αυτό, το υποστηρίζω, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να αποφύγουμε ε, διπλές αμοιβέ, κάτι το οποίο θα ήταν αντιπαραγωγικό και μιλάω κυρίως για ε, τέλη αφού γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι υπερβολική η αμοιβή, το τέλος που θα ε, χρεωθεί, κάτι το οποίο μπορεί να είναι κακό για τους δημιουργούς. Η ιδέα τώρα της, ε, του επιπλέον τέλους για τα έργα τα οποία θεωρούνται έργα που αποσκοπούν σε ένα συγκεκριμένο κοινό, ε, κατά τη γνώμη μου, Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο είδους ανταμεφή ε, σε σχέση με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, τους παραδοσιακούς ε, εφόσον θα ε, δώσουμε, θα, η διαδικασία ε, αδειών θα είναι πλέον πολύ πιο ε, δαπανηρή, κάτι το, το οποίο σημαίνει ότι θα είναι πολύ πιο ευάλωτη η θέση όλων αυτών των δημιουργών εις βάρος της ευρωπαϊκής ποικιλομορφίας που κατάλαβα ότι θέλετε να την υποστηρίξετε. Αν θέλετε όμως να το κάνετε αυτό, δεν πρέπει να ε, κάνετε μία, ε, ένα περιορισμό στο 30%. Φαντάζεστε ότι μόνο 30% ε, ευρωπαϊκές ταινίες προβάλλονται στην Αμερική, για παράδειγμα, ή στο διαδίκτυο. Πρέπει πραγματικά να δούμε τα πράγματα κάπως πιο ισότιμα, για να μπορέσουμε δηλαδή να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας, αλλά να μην αντιταχθούμε και στον εξυγχρονισμό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γκεργέρο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω κάποια σύντομα σχόλια για το σχέδιο κειμένου. Πρώτα-πρώτα με μεγάλη μας ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι ο πύχη είναι αρκετά ψηλά όσον αφορά την αρχή της χώρας προέλευσης. Ήταν ψηλά και έμεινε ψηλά. Έχουν γίνει κάποιες μεταβολές, αλλά αντιλαμβανόμεθα ότι ο εισαγωγής θέλησε έτσι να διαμορφώσει τις προτάσεις μας και Βεβαίω αυτή ε, η προβληματική έχει δυσκολίε. Καταλαβαίνουμε ποιε είναι οι ανησυχίε όπω διατυπώθηκαν για ειδικά αυτό το σημείο. Πάντω θα πρέπει να θυμηθούμε τα όσα ήδη έχουμε συζητήσει. Θα συνεχίσουμε πάντως να το συζητούμε και για άλλη μια φορά εμείς εμένουμε στην άποψη ότι η πρότασή μας διατυπώνει αυτή την αρχή με τρόπο αυστηρά περιχαρακωμένο όσον αφορά αυτές τις ε, πρόσθετες πληρωματικές υπηρεσίες από πλευρά του παρόχου. Τα λέμε και στις αιτιολογικές διατάξεις προτασής μας και λέμε ότι η συμβατική ελευθερία δεν θίγεται, η ελευθερία των συμβάσεων τέλο πάντων. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση που απορρέει από τον κανονισμό αυτό, ούτω ώστε υπάρχει να παρέχουν ε, τέτοιες ευρείες και διασυνοριακές υπηρεσίες. Ελπίζουμε δε ότι το αποτέλεσμα θα είναι να υπάρχει ευρύτερη διαθεσιμότητα όλων αυτών των προϊόντων και μορφών περιεχομένου. Πάντως μία υποχρέωση δεν επιβάλλουμε το κείμενό μας, την πρότασή μας. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση του εισηγητή, συμφωνούμε με κάποια από τα όσα αναφέρθηκαν. Ιδίως αυτή η περιγραφή των υπηρεσιών που στοχεύουν σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ότι αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει αναγκαστικά να επιβληθεί. Το συζητήσαμε κατά συνέχιση του κειμένου μας και καταλήξαμε στο ότι η πιθανότητα επανεγκατάστασης του παρόχου ούτως ώστε να αναζητήσει πιο ευεργητικές ε, και ευμενείς διατάξεις ε, είναι κάτι το οποίο δεν θα συμβεί και αν συμβεί τέλο πάντων θα είναι σπάνιο. Επίσης, σε αυτό το σημείο ληφθεί υπόψη ότι για τον ελόγο κανονισμό δεν κινούμεθα στα πλαίσια του διοικητικού δικαίου των εθνικών των κρατών μελών αλλά κινούμεθα στα πλαίσια του δικαίου πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού. Ε, γι' αυτό σας λέω, δεν υπάρχει ουσιαστικό κίνδυνος ε, μετακίνησης των παρόχων από χώρα σε χώρα. σάγρα ευμενέστερου νόμου. Τώρα έχουμε κάποιες και νέες προτάσεις, ούτως ώστε να δούμε τι είδους διαφορετικές ρυθμίσεις θα ισχύσουν όσον αφορά την αμοιβή, ανταμοιβή, ε, δημιουργών και συμφωνούμε. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δίκαιη ανταμοιβή. Για κάθε περίπτωση ιντερνετικής μετάδοσης. Αλλά θέλουμε ότι αυτό πρέπει να ρυθμιστεί στον ερωδοκανισμό. Αλλά στην οδηγία για το copyright και την ενιαία αγορά. εκρεμεί η συζήτησή τη εδώ στην Επιτροπή σας και εκεί έχουμε μια σειρά άρθρων που έχουμε συντάξει ούτω ώστε να θωρακίσουμε τους, τα δικαιώματα των δημιουργών και να βελτιώσει η θέση τους όσον αφορά την αμοιβή που δικαιούνται. Προσοχή επίσης όσον αφορά τη θέσπιση μηχανισμού δύναμη του οποίου η αδειοδότηση αφορά κάποια δικαιώματα κάποια δικαιώματα τα οποία τώρα θα είναι πιο δύσκολο να ασκηθούν από πλευρά κρατικών και μη ε, παρόχων λόγω της δημιουργίας συμπληρωματικών δικαιωμάτων κοντά σε εκείνα. Επίσης για τις αναμεταδόσεις ασχολείται εν μέρη και με αυτό ο κανονισμός θα πρέπει βεβαίω και να μελετηθούν πιο προσεκτικά αυτές οι διατάξεις και σημειώνουμε ότι η καλωδιακή μετάδοση αποτελεί κάποια παροχή υπηρεσιών και η προτινόμενη νέα ε, μετάδοση με τον τρόπο injection έχει αποτελέσει αντίγυμνο νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Direct injection. Πρόκειται για μέθοδο που συζητείτε και άρα θα πρέπει να το κοιτάξουμε πιο προσεκτικά. Αυτά και ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Επρόκειται και το σημείο υπαριθμών 4, δεν βλέπω άλλος να ζητεί το λόγο επ' αυτού και σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η πέμπτη 22 έκτου. Φέτος βέβαια, το μεσημέρι. Συνεχίζουμε. Σημείο παραθμόν 5. Συζήτηση ε, τη έκθεση για την καταπολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε μέσω του ποινικού δικαίου. Το λόγο και ο κ. Χρυσόγονο που είναι ο Πρόεδρε, ευχαριστώ. Οι πρόσφατε τρομοκρατικέ επιθέσει στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ανέδειξαν την ανάγκη ότι θα πρέπει να προλαμβάνουμε αλλά και να τα την τρομοκρατία. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται με όσο γίνεται πιο αποτελεσματική χρήση των καταλήλων μέσων. Άρα θα πρέπει να κόψουμε τη χρηματοδότηση αυτών των τρομοκρατικών ε, συμμοριών και έτσι θα μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Και θα χρειάζεται μέσα από αποτελεσματική νομοθεσία για ε, το ξέπλυμα χρήματος και έτσι θα περιορίσουμε και τη φοροδιαφυγή και το οργανωμένο έγκλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα σχετικά νομοθετικά μέσα. Έχουμε τη σχετική ποινική νομοθεσία, το θέμα της συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών αρχών, ούτω ώστε υπάρχουν και οι διαδικασίες συνταλλαγής πληροφοριών, υπάρχει επίσης η νομοθεσία πρόληψης και καταπολέμησης της διάθεσης προϊόντων εγκλήματος και την νομιμοποίησή τους και οπότε αυτό το κείμενο, όπως λέει και ο τίτλος του, έχει ως στόχο να βελτιώσει την χρήση των εν μέσων. Θεωρούμε ότι η πρόταση πετυχαίνει το στόχο της με εφαρμογή και υλοποίηση των διεθνών υποχρεώσεών μας επί τη βάση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά την ε, κατάσχεση, τη δίμευση, την έρευνα ε, και επίσης τα έσοδα από το έγκλημα και έχουμε επίσης και κάποιες σχετικές συστάσεις που προέρχονται από την Task Force Financial Action, FATF. Θεωρούμε ότι είναι εύστοχα όσο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως θα πρέπει σε κάποια σημεία να προβληματιστούμε λίγο παραπάνω και θα πρέπει επίσης να προσέξουμε ιδιαίτερα το θέμα της διαφάνειας του ανοιχτού πνεύματος όσον αφορά το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να διευκολύνουμε τις σχετικές προσπάθειες τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν κάποιο είδους μητρώα για κάθε δικαιούχο νομικού προσώπου ή ιδρύματος. Οπότε το αν, το ξέρουμε ακριβώ είναι ο δικαιούχο κάθε φορά, ο πραγματικό δικαιούχο, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, ώστε να έχουμε την πρόληψη αλλά και την καταστολή του εγκλήματος. Και οι αρμόδιες αρχές που εποπτεύουν ε, το πώς λειτουργούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με αυτή την οδηγία θα πρέπει να μπορούν να ανταλλάξουν εμπιστευτικές πληροφορίες άσχετα με το ακριβές περιεχόμενο ή τη φύση κάθε υπηρεσία. Θα πρέπει να βρούμε βέβαια τη σωστή νομική βάση για αυτή τη δυνατότητα έλεγχη πληροφοριών διαβαθμισμένων. Και έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται όσον αφορά τα όσα διεθνώ ισχύουν. Οι πληροφορίες φορολογικές, ε, τα μητρώα σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, θα πρέπει και αυτά να βοηθούν την ανταλλαγή πληροφορία μεταξύ φορολογικών αρχών και των άλλων συναρμοδίων κανονιστικών και δίπλικων αρχών. Πληροφορίες σε σχέση με καταπολέμηση της ε, οικονομικής τρομοκρατίας αλλά και ξεπλήματος ε, χρήματος θα πρέπει να αποτελεί επίσης αντικείμενο εποπτείας από, αυτές, του αυτούς τους φορείς. Άρα, ανταλλαγή πληροφοριών, συνεργασία όλων αυτών των αρμοδίων αρχών, αλλά και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Χρειάζεται επίσης και εποπτεία. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται απαρακόλλητα. Έστω και ακούσια με κάποιο είδου απουσία ασφάλεια δικαίου. Που προκύπτει όταν δεν υπάρχουν ρητέ διατάξει που τα ρυθμίζουν όλα αυτά. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το νομικό πλαίσιο που είναι ακόμα πιο σημαντικό. Μια που αυτού του είδου η εποπτεία σε πολλέ περιπτώσει ασκείται από κάποιες αρχές που δεν ασχολούνται με το ξύλιμα χρήματος, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα. Επίσης, να τονίσουμε ότι τα εθνικά δεδομένα, τα σχετικά με τον εντοπισμό κάποιων ε, λογαριασμών και κάποιων θηρίδων τραπεζικών που ανήκουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο, τώρα ε, είναι κάτι το οποίο γνωρίζει κατάτμιση Γιατί δεν μπορούν όλα αυτά να αξιοποιηθούν από τις υπηρεσίες πληροφοριών και των άλλων συναρμοδίων υπηρεσιών εγκαίρως. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάποιο είδους κεντροκατευθυνόμενους μηχανισμούς όπως κάποιο μητρέο, ένα σύστημα ανταλλαγή ε, πληροφοριών κοινό στα κράτη-μέλη και έτσι αποτελεσματικά και έγκαιρα να υπάρχουν πληροφορίε όσον αφορά την ταυτότητα των δικαιούχων κάποιων τραπεζικών λογαριασμών και των ε, ιδιοκτητών κάποιων ε, θηρίδων τραπεζών και των πληροξουσίων τους κλπ. κλπ. βέβαια υπάρχει το θέμα του επαγγελματικού απορρίτου, υπάρχει το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίγη και Παρακαλούμε, μιλήστε πιο αργά για να μεταφράσετε ευκολότερα, λέει ο πρόεδρο, τον κύριο Χρυσόγονο. Υπάρχει επομένω το θέμα επαγγελματικού απορρίτου, το θέμα του δικαιώματο στον ιδιωτικό βίο και το δικαίωμα σε δίκη, δίκη. Όλα αυτά θα πρέπει να φύγονται από την συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών ή από κάποιες συνήθεις ε, συναλλαγές επί τη βάση απλών υποψιών. Οπότε για να αντιμετωπιστεί το ξέπλυμα χρήματο αποτελεσματικά, επιτακτικό είναι τα χρηματοπιστωτικά κέντρα, τα υπεράκτια ή μη υπεράκτια ή η φορολογική παράδειση να μην επιτρέπεται να προβαίνουν σε επιδιαιτησία κανονιστικού ή άλλου είδους σε κάποιες ε, παράνομες αγιαθέμπτες συναλλαγές που οδηγούν σε φοραπαλλαγή και φοροδιαφυγή. Αυτά τα υπεράκτια κέντρα θα πρέπει να αποσυνδεθούν από το οικονομικό και το πιστοτικό γίγνεσθε της Ένωσης. Οπότε θα πρέπει να έχουμε κάποια καλά σταθμισμένα μέτρα για το ξέπλυμα και έτσι να προστατεύονται τα συμφέροντα τα οποία φύγονται από το οργανωμένο έγκλημα. Χρειάζονται επομένω δικαστικέ, νομοθετικέ προσπάθειε. στόχο ναι, να έχουμε όσο γίνεται πιο πολύ ασφάλεια δικαίου. Και ταυτόχρονα να σεβόμεθα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η δε προθεσμία για τις τροπολογίε στον σοβαρό κείμενο είναι η 8η έκτου ενεστώτος έτους το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φώσος. Εγώ αντικαθιστώ την σκιώδη συγγήτριά μας την κυρία Ράντερ, γι' αυτό και θα ήθελα να παρουσιάσω τις προτάσεις και τις απόψεις Τα τελευταία τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενδυναμώσει τα μέτρα ασφάλειας, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, όλα αυτά για να δημιουργηθεί μια πιο ασφαλής Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση αυτή είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί θα επιτρέψει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διοκτικών αρχών, των κρατών μελών και των αρχών αυτών που καταπολεμούν την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει αντίστοιχη οδηγία η οποία είναι υπό τροποποίηση. Γι' αυτό και θα πρέπει να προσέξουμε πού θα στοχεύσουμε τις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρουζιέρα, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη γνωμοδότησή του. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση που ουσιαστικά θα ενισχύσει τα όπλα που διαθέτουμε για να καταπολεμήσουμε την εγκληματική αυτή δραστηριότητα που στηρίζει και χρηματοδοτεί εν μέρη και την ε, τρομοκρατία. Πρόκειται για 3,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ και για κάποια κράτη-μέλη συγκεκριμένα έχουμε ενδείξεις που δείχνουν ότι ο διασυνοριακός χαρακτήρας αυτού του οργανωμένου εγκλήματος μπορεί να φτάνει μέχρι και το 50% των διαπιστωμένων εγκληματικών πράξεων που αναφέρονται σε αυτή την κατηγορία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε για τον καθορισμό της νομοποίησης ε, εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, τον ορισμό, η πρόταση της ε, Επιτροπής έχει σαν σκοπό να μας οδηγήσει σε μια αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση. Οι προτάσεις αυτές συμπληρώνονται πολύ σωστά λοιπόν με αυτές τις ε, ιδέες που μόλις ακούσαμε όσον αφορά την κωδικοποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων σε σχέση με την ε, σύμβαση της Βαρσοβίας και άλλους διεθνείς ε, ε, υποχρεώσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ θετικό. Επίσης, οι υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαφάνεια για τους τελικούς δικαιούχους. Αυτή η διαφάνεια είναι απαραίτητη όσον αφορά τη νομιμοποίηση κάποιων εσόδων ο τελικός δικαιούχος και η διαφάνεια όσον αφορά τους τελικούς δικαιούχους είναι κάτι το καθοριστικό. Θα πρέπει να επιλέξουμε τον καλύτερο τρόπο για να φτάσουμε σε αυτήν τον εντοπισμό, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Καθοριστικό είναι επίσης να υπάρχει πραγματική ανταλλαγή πληροφοριών για να λειτουργήσουν σωστά οι πληροφορίες. Στηρίζω λοιπόν την πρόταση του εισηγητή και βεβαίως και η αναφορά στον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που επίσης είναι σημαντική διευκρίνηση. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την υποστήριξή του για την πρόταση. Όπως επίσης ανέλαβε το θέμα αυτό και το εξετέλεσε με μεγάλη ταχύτητα. Ε, στη, στο Συμβούλιο επίσης ε, φτάνουμε σε μια γενική προσέγγιση και θέλουμε αυτή η πρόταση να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν. Όσον αφορά την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου, η πρόταση σκοπό έχει να συμπληρώσει την οδηγία για την ε, καταπολέμηση νομοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ε, θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τα θέματα αυτά ήδη καλύπτονται από τη σχετική οδηγία και καλό είναι να μην τα ξαναναφέρουμε εδώ για να αποφεύγεται σύγχυση. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ για αυτή τη σύντομη παρατηρήση. Δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Παρακαλώ, λοιπόν, σημειώστε ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 8η Ιουνίου. 8 Ιουνίου, λοιπόν, ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο, το 5 της ημερήσιας διάταξης και συνεχίζουμε με το σημείο 6, ανταλλαγή απόψεων για το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ο λόγος τον κύριο Φως, που είναι και ο εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ πρόκειται για την πρόταση της Επιτροπής. Έχω μείνει άναυδος να σας πω, με αυτά που μας έχει υποβάλει η Επιτροπή. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω, γιατί είναι κάτι μεταξύ ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ε, προστασίας δεδομένων και τελικά ποιοι είναι οι στόχοι που έχουμε θέσει για την εσωτερική αγορά. Ανάπτυξη, στήριξη της οικονομίας, της ευρωπαϊκής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Πρόκειται λοιπόν για ροή δεδομένων που με κανένα ε, τρόπο δεν πρόκειται να επιτευχθούν. Δεν βλέπω να υπάρχει στόχος ε, που να μας οδηγεί στο μέλλον. Εδώ βλέπουμε την DG Connect, την DG Justice, οι οποίες ενδεχομένως έχουν ενδιαφέρον ε, σε αυτό το θέμα, αλλά πρόκειται για μία πρόταση που αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη. Καλό θα ήταν η Επιτροπή να μας έλεγε ε, διατηρήστε τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των ε, δεδομένων των πελατών σας, προσπαθήστε να μην παραβιάσετε τις αρχές ε, που εμπεριέχονται στο χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φτάνει. Κοιτάξτε, έχουμε πάρει αποφάσεις για τα θέματα αυτά, οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί και γι' αυτό και αναφέρομαι σε αυτά που θα έπρεπε να είχαν γίνει και βλέπουμε την Επιτροπή να μας προτείνει εδώ μια πολύ εξειδικευμένη νομοθεσία. Δηλαδή, είναι σαν να αγνοούμε έναν κανονισμό, τον οποίο συζητούμε εδώ και πέντε χρόνια, για τον οποίο υπήρξε επεξεργασία, διαπραγμάτευση και ξαφνικά υπάρχει μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη. Ακόμα και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι πολύ περίεργες. Η προστασία των δεδομένων, το αντικείμενο ε, του συγκεκριμένου κανονισμού, μπορεί κανείς να πει ότι πρέπει να συμπληρωθεί, αλλά δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε εδώ ένα νέο καθεστώς, να ε, δημιουργήσουμε από το μηδέν ένα νέο καθεστώς για το ίδιο θέμα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να στηριχτούν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μην υπάρχει δηλαδή ένας μονοπωλιακός χειρισμός και επεξεργασία των δεδομένων. Μα ακριβώς το αντίθετο όμως πετυχαίνουμε αν ακολουθήσουμε τις προτάσεις αυτές της Επιτροπής. Δηλαδή οι μεγάλοι, οι πολυεθνικές, οι μεγάλοι όμιλοι, έτσι και αλλιώς αυτή τη στιγμή είναι παντοδύναμες. Τους δίνουμε ακόμα περισσότερα δικαιώματα. Είναι πάρα πολύ απογοητευτικό αυτό που βλέπω εδώ και σε καμία περίπτωση δεν νομίζω ότι μπορούμε να την τροποποιήσουμε την πρόταση αυτή για να γίνει κάτι το επικοδομητικό και θετικό. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι στόχοι που θα έπρεπε να μας οδηγήσουν προς περισσότερη ανάπτυξη. Όντως λείπουν κάποιες κωδικοποιήσεις, κάποιες ε, τροποποιήσεις, θα πρέπει κάποιες τεχνολογίες να ενσωματωθούν. Υπάρχουν κάποιες μικρές προτάσεις που ενδεχομένως θα μπορούσα να τις δεχτώ, αλλά η λεγόμενη επικοινωνία με τους ε, λεγόμενους OTTs βεβαίως είναι κάτι που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, αλλά σε καμία περίπτωση τίποτα περισσότερο. Να σκεφτούμε ε, την επικοινωνία αλλά οι επιπτώσεις μιας τέτοιας πρότασης είναι σαν να μην λαμβάνονται καθόλου υπόψη. Πραγματικά λοιπόν, από τη μία υπάρχει επικάλυψη με την ε, υπάρχουσα νομοθεσία και αναρωτιέμαι πώς μπορεί κάποιος να κατανοήσει τι κάνει εδώ η Επιτροπή από τη στιγμή που τα ίδια πράγματα εμπίπτουν και στον ένα κανονισμό και στη νέα πρόταση κανονισμού. Μα αν υπάρχουν παραβιάσεις, θα υπάρχουν δύο συστήματα κυρώσεων. Δεν καταλαβαίνω, επαναλαμβάνω, υπάρχει συγκεκριμένη επικάλυψη. Τι θα κάνουμε με τις παραβιάσεις, τι θα κάνουμε με τις ε, κυρώσεις, τι θα κάνουμε με την άμεση διάθεση στην αγορά, με την άμεση εμπορευματοποίηση, τι θα κάνουμε με τις άδειε. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουμε απολύτω καμία συνοχή και πιστεύω ότι θα προκαλέσουν μεγαλύτερη σύγχυση εάν ποτέ υιοθετηθούν. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν πιστεύω ότι εδώ πρέπει να κοιτάξουμε μόνο τα μεταδεδομένα. Κάτι που είναι συμπληρωματικό με τον υπάρχοντο κανονισμό και να δούμε ποιο είναι ο πιο σωστό τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα μεταδεδομένα. Επίση, κάποιοι ορισμοί, το θέμα τη επικοινωνία, όπω σα είπα, έχουμε τον ε, Ευρωπαϊκό Κώδικα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και εδώ όμως δεν υπάρχει καμία συνοχή στους ορισμούς. Έχω την εντύπωση ότι δεν κοιτάμε προς το ψηφιακό μέλλον. Και υπάρχει σήμερα μια τέτοια πληθώρα προσφορών και δυνατοτήτων που έχω την εντύπωση ότι έχουμε τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ε, εμπιστευτικά δεδομένα και όλες αυτές οι κατηγορίες είναι σαν να μην υπάρχουν. Οι ορισμοί δεν λαμβάνουν υπόψη τους εδώ αυτές τις διαφοροποίησεις. Για το θέμα των cookies. Τα first party και τα third party cookies. Και ε, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει καλύτερα αν πραγματικά υπάρχει κίνδυνος για τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε, αυτά, σε αυτές τις κατηγορίες ε, των cookies. Νομίζω όμως ότι τελικά οδηγούμαστε προς μία κατάσταση όπου θα υπάρχουν μόνο first party cookies και ότι όλα τα δεδομένα αυτά θα βρίσκονται μέσα στους browser. Ήδη μεγάλες επιχειρήσεις από ό,τι ξέρω αυτό κάνουν. Προ τα εκεί λοιπόν πάει η τεχνολογία. Άρα και αυτή η πρόταση δεν είναι χρήσιμη. Τώρα, όσον αφορά τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, εγώ που είμαι μία μικρή ε, επιχείρηση, μία μικρομεσαία επιχείρηση, είμαι πάροχος πληροφοριών και επικοινωνίας, πού γίνεται η κατηγοριοποίηση και πού υπάρχει διαχωριστική γραμμή. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι και σε αυτό το τομέα η, τα μέτρα ασφάλειας, η εμπιστευτικότητα, οι διαχωριστικές γραμμές δεν έχουν τεθεί με σκοπό ο χρήστης να γνωρίζει αν το δίκτυο το οποίο χρησιμοποιεί είναι ασφαλές ή όχι. Και αν με τα μέτρα αυτά αυξάνεται η ασφάλεια. Έχω και άλλα σημεία που θα μπορούσα να σας τα παρουσιάσω αν είχαμε το χρόνο και αν επιθυμούσατε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πλειοψηφία. Α, εν πάση καταλάβατε ποιο είναι το γενικότερο μήνυμα. Να αναφερθώ συγκεκριμένα στο άρθρο 4 της πρότασης κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Επικοινωνιών. Εδώ ενδεχομένως θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, αλλά στο σχέδιο προτάσεων δεν γίνεται απολύτως καμία διάκριση μεταξύ δεδομένων περιεχομένου πληροφοριών. Πρόκειται για μια πολύ γενική διατύπωση και πιστεύω ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη από του περιεχομένου εδώ και καλύτερη διατύπωση. Αναφερόμαστε λοιπόν στην ψηφιακή επικοινωνία και απόρριτα δεδομένα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Παραδείγματο χάρη, φαντάζομαι ότι εδώ συμπεριλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ ενό νοσοκομείου που ενδεχομένω μπορεί να μεταδώσουν κάποια προσωπικά δεδομένα που αφορούν του ασθενεί, ιατρικού φακέλου. Ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της ψηφιακής μετάδοσης. Έχω την εντύπωση ότι και εδώ χρειάζεται πιο συγκεκριμένη διατύπωση. Είμαι λοιπόν πάρα πάρα πολύ επιφυλακτικός, νομίζω το καταλάβατε. Υπάρχει θέμα συνοχής. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει ένας κανονισμός για την προστασία των δεδομένων, ίσως θα μπορούσαμε να βασιστούμε σε αυτό και ενδεχομένως να συμπληρώσουμε με κάποια επιπλέον μέτρα. Δεν πιστεύω ότι οι στόχοι είναι ξεκάθαροι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ξέρει τι αποφασίζει και με ποιο τρόπο θέλει να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτή η πρόταση δεν κοιτάει το μέλλον και σε καμία περίπτωση δεν αποφεύγει τις επικαλύψεις. Ευχαριστώ πολύ κύριος Νεγκρέσκου. Συγγνώμη, περίμενα να τελειώσει η διερμηνία στα αυτιά μου Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη για το συγκεκριμένο κείμενο. Συμφωνώ ε, με κάποια από τα στοιχεία που τόνισε ο κύριος Φως. Ε, είναι για μας πολύ σημαντικό τους για μας τους Ευρωβουλευτές να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών μας. Όμως μου φαίνεται ότι αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντί να κάνει κάτι για τους πολίτες ε, έγινε για να καταπολεμήσει κάτι και κάνοντας το αυτό δημιούργησε κάποια προβλήματα. Κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα ξεκινά από την ιδέα ότι ο διαχειριστή των δεδομένων είναι ήδη ένοχο για κάτι. Δηλαδή, το τεκμήριο τη αθωότητας θα έπρεπε να υπάρχει κάπω μέσα σε αυτόν τον κανονισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ξέρετε, όπω έχει τονιστεί και προηγουμένω. Ε, υπάρχει ο κανονισμό γενικό για την προστασία των δεδομένων που ε, ορίζει πώς πρέπει να γίνει η διαχείριση των δεδομένων και εμείς ήδη δυσκολευτήκαμε να συμφωνήσουμε από αυτού του κανονισμού. Ανοίγουμε λοιπόν και πάλι το κουτί της Πανδώρας τώρα και ξέρουμε ότι για τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων υπάρχουν ακόμη κάποια περιθώρια ερμηνεία διαφορετικά και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό ο κανονισμό σε εθνικό επίπεδο να εφαρμοστεί. Για να επανέλθω λοιπόν, ε, γιατί εντάξει, πρέπει να εξετάσουμε την πρόταση αυτή. Αν μιλούμε για ζητήματα ιδιωτικής ε, ζωής ε, πρέπει να σκεφτόμαστε και την παρέμβαση ε, λόγω του hacking, λόγω ε, κάποιων κρατικών μηχανισμών. Δεν μιλάμε, νομίζω, δεν αναφέρεται παρκώς αυτό στον στην έκθεση. Μιλούμε επίσης για την κυριότητα των δεδομένων και αυτό δεν ορίζεται επαρκώς. Έχουμε νομίζω πάντως κάποιο συμβιβασμό σε σχέση με τον ορισμό αυτού, αυτής της κυριότητας των δεδομένων. Κάτι ακόμη, ακόμη. κάθε φορά πρέπει να ζητούμε καλύτερη ψηφιακή εκπαίδευση. Πάντοτε μιλάμε για την προστασία τη ιδιωτική ζωή και των ε, προσωπικών δεδομένων, όμω η πληροφορία παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Πρέπει να ζητούμε από όσου χρησιμοποιούν πολλά από τα δεδομένα μα, να ενημερώνουν καλύτερα του πολίτε. Ε, αυτό πρέπει να γίνεται βέβαια πραγματικά, όχι να κάνει προς κλικ ε, στην αποδοχή κάποιων όρων και κανεί δεν του διαβάζει. Πρέπει κανεί όντω να παρέχει την πληροφόρηση αυτή και να κάνει πολύ περισσότερα και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να προκύψει από εμά, να είναι μια δική μας συμβολή σε αυτήν την κοινή συμφωνία. Τώρα, η κωδικοποίηση. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε εδώ, γιατί στο έγγραφο αυτό ε, υπάρχουν, νομίζω, υπάρχει απουσία πολλών τεχνικών στοιχείων και τεχνική προσέγγιση. Εγώ προέρχομαι από τον ψηφιακό τομέα, δουλεύω σε αυτό το τομέα και όταν βλέπω καμιά φορά έναν κανονισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν δεν, το βλέπω ότι δεν καταλαβαίνουν πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Ξεχνούν στην πράξη πώς θα εφαρμοστούν όλοι αυτοί οι κανονισμοί τους οποίους προτείνουν. Το βλέπω για παράδειγμα και στα συγκεκριμένα άρθρα, τα οποία, ε, πολλά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν, ενώ υπάρχουν λύσεις που μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν. Πρέπει και αυτό να το λάβουν υπόψη λοιπόν και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ε, για τις τεχνικές πτυχές των προτάσεων που υποβάλλουν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντελβού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι όλος ιδιαίτερος ε, που συνεργάζομαι ως και συγγήτρια με τον κύριο Φως ε, μετά από αυτήν την παρέμβασή του που ήταν τόσο ένθερμη, με τόσο ζήλο. Σπανίως τον έχω ακούσει τόσο αποφασισμένο για ένα ζήτημα ε, όσο σήμερα και νομίζω ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη συζήτηση, όχι μόνο εδώ στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, αλλά και εντό των πολιτικών ομάδων, γιατί πρέπει να καταλήξουμε σε θέσεις ε, οι οποίες να είναι κάπως ευθυγραμμισμένες. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να ε, λύσουμε το πρόβλημα της εμπιστευτικότητας, γιατί όλοι θέλουμε ε, οι επικοινωνίες μας να είναι προστατευμένες και εμπιστευτικές. Αυτό είναι κάτι ε, για το οποίο συμφωνούμε, τουλάχιστον επ' αυτού συμφωνούμε. Και πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ε, την συνοχή μεταξύ των διαφόρων οδηγιών και κανονισμών ε, που ε, έχουμε εγκρίνει και τις οποίες πρόκειται να εγκρίνουμε ή τις οποίες επεξεργαζόμαστε. Είναι ο ρόλος της δικής μας Επιτροπής να εξετάζουμε ότι υπάρχει αυτή η συνοχή μεταξύ του ενός κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα, ε, της οδηγίας ε, για τις ψηφιακές επικοινωνίες. Εγώ χαίρομαι πολύ που ε, εργάζομαι επί του θέματος αυτού και πρέπει να σας ομολογήσω ότι η δική μου προσωπική άποψη δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως ακόμη. Έχω ακόμη πολλές αμφιβολίες, πολλά ερωτηματικά και πιστεύω συνεπώς ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εργασία και πολύ συναρπαστική. Αλλά νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ποιο θα είναι το θετικό αποτέλεσμα αυτό, εγώ αναρωτιέμαι πάντως. Κύριε Άντερσον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι προφανές ε, ότι αυτό, ε, αυτή η εργασία θα είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ε, εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέτει αυτό το ζήτημα και που υπέβαλε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Η άποψή μου επί της προτάσεως αυτής είναι ότι δεν είναι αρκετά ισχυρή ως προς την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των, δεδομένων, ε, των προσωπικών δεδομένων επικοινωνίας. Υπάρχουν κάποια δύσκολα θέματα ε, επί των οποίων πρέπει να εξευρεθεί μια ισορροπία. Αυτό θα είναι κάτι ε, το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε πολύ λεπτομερώς στην, μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Υπήρξε μία προηγούμενη εκδοχή ε, του θέματος αυτού που μας υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτερη εκείνη η εκδοχή. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να αποκατασταθεί αυτή η προηγούμενη εκδοχή. Παράδειγμα, η ιδιωτική ε, ζωή ε, που να μην ε, αποτελεί, να, να μην είναι απλώς εναλλακτική ε, επιλογή, να είναι υποχρέωση. Νομίζω ότι ήδη έχουμε αναθεωρήσει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και κάποια ζητήματα καλύπτονται και από την οδηγία του e-privacy, της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο, ε, το 2002 θυμάμαι. Προϊστορία είναι πλέον αυτό. Είναι καλό λοιπόν να αναθεωρηθεί αυτή η οδηγία και να καταστεί κανονισμός. Κάτι πρέπει να γίνει, νομίζω. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή κατά πόσο θεωρεί ότι είναι αποδεκτή λύση να υπάρχει ένα συνδυασμός του κανονισμού προστασίας δεδομένων και της οδηγίας e-privacy. Θεωρείτε ότι θα ήταν καλό αυτό και για τους χρήστες και για τις εταιρείες. Ε, δεν ξέρω, αυτό εννοούσατε. Εντάξει, μπορεί να είναι η υπερβολή αυτό ε, που είπα, αν βλέπω καλά από την αντίδρασή σας και από το ότι ανασηκώνετε το φρύδι σας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπορέσουμε να αναθεωρήσουμε και τα δύο νομοθετήματα, να αρχίσουν να ισχύουν ε, οι δύο νομοθεσίες συγχρόνως, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα ε, ερμηνείας της νομοθεσίας αυτής και εφαρμογής της. Κάτι ακόμη. Ε, κατά πόσο θα έπρεπε να αναφέρεται το θέμα της, των ε, ε, λόγων για τους οποίους θέλουμε να ε, λαμβάνεται τόσο υπόψη η ιδιωτική ζωή αυτή. Τώρα το θέμα του cookie fatigue, δηλαδή η υπερβολική ύπαρξη των cookies, όλη την ώρα εμφανίζονται αυτά τα cookies που πρέπει να τα αποδεχθούμε και όλος ο κόσμος θεωρεί ότι η ιδιωτική του ζωή παραβιάζεται επειδή όλο και περισσότερα cookies εμφανίζονται. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Τώρα, πώ θα το κάνουμε αυτό, θα βρούμε μια ισορροπία, πρέπει να το σκεφτούμε, θα δούμε πώ θα το κάνουμε, αλλά σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα, το θέμα του του tracking wars, Τον tracking wars. Δεν ε, μπορεί κάποιος ε, να διαβάσει έναν ιστότοπο αν δεν αποδεχθεί τα cookies Εμένα δεν μου αρέσει αυτό, ειδικότερα ως προς τους δημόσιους ιστότοπους που χρηματοδοτούνται από δημόσιο χρήμα και γι' αυτό κάτι πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα μπορεί να βρεθεί μια συνένεση και ως προς αυτό. Τώρα, το online και το offline tracking, όταν δηλαδή γίνεται κάποια, κάποιος εντοπισμός, ακόμη και αν κάποιος δεν χρησιμοποιεί ένα δίκτυο, αυτό είναι κάτι, ε, δεν είναι κάποιος έναν ιστότοπο, αυτό ε, νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα που επίσης πρέπει να λύσουμε. Είμαι βέβαιος ότι θα το συζητήσουμε πάρα πολύ αυτό στο μέλλον και πραγματικά προσδοκώ τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ. Ε, εμείς ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε μείνει πολύ πίσω στο το χρονοδιάγραμμα γιατί έχουμε άλλα τρία θέματα να συζητήσουμε που είναι πολύ σημαντικά και για αυτά τα τρία έχουμε 30 λεπτά. Δεν έχει δει κάποιο άλλο το λόγο για το συζητούμενο θέμα, το υπαριθμό 6, οπότε και συνεχίζουμε με το 8. 8 λοιπόν εννοεί το 7. Όχι, το 8. Μέτρα προστασία των καταγγελόντων που ενεργούν προ το δημόσιο συμφέρον κλπ. Δώσουμε το λόγο η στην εισηγητρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι μπορούμε τώρα να συζητήσουμε έτσι αυτό το θέμα γιατί έμεσα ή άμεσα μας έχει εμπνεύσει στα τρία πρώτα χρόνια αυτής της ε, θητείας. Είχαμε το Lux Leaks, το σκάνδαλο, είχαμε γενικότερα το θέμα του ότι θα πρέπει να δίνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για να προστατεύονται τα θεμητά συμφέροντα των Ευρωπαίων. Όλα αυτά επομένω αγγίζουν πάρα πολύ τι συζητήσει μα και επίση όλα αυτά τα έχουμε ήδη συζητήσει και ασχολήθηκε με αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πρωτοβουλία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σχετική προστασία που θα πρέπει να θεσπιστεί, να είναι ευρύτερη, ε, είναι κάτι το απαραίτητο για αυτού τους καταγγέλλοντες. Και στα διάφορα κράτη-μέλη η κατάσταση είναι πολύ ανομοιογενής. Έχουμε τελείως διαφορετικές ρυθμίσεις. Έχουμε τώρα έξι κράτη-μέλη που προβλέπουν προστασία για τους καταγγέλλοντες. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι όμως τόσο λειτουργική. Το Λουξεμβούργο έχει κάποιο είδους ε, προστασία, αλλά δεν εμπόδισε αυτό από το να καταδικαστούν αυτοί που κατήγγυλαν τα του Λιξ. Πάντως υπάρχει ευρεία συνένεση. Πρέπει του καταγγείλτες να του προστατεύσουμε. Και επομένω αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Θα επικαλεστούμε την κείμενη νομοθεσία του, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Δικαστηρίου τέλος πάντων, όσον αφορά την προστασία του δημοσίου συμφέροντο. Πολύ σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση και Θέλω να προβληματιστούμε, συνάδελφοι και ιδίω οι σιωδησηγητές, κάποια στοιχεία αυτά θα πρέπει να μας βοηθήσουν. Πώς ορίζεται ένας καταγγέλων. Δύο είναι οι στόχοι. Σε ποια περίπτωση έχουμε καταγγελία. Να έχουμε έναν ευρύ ορισμό. Ε, μισθωτός, είναι εμπειρογρόμων, είναι υπάλληλο, ε, μπορεί να είναι εξωτερικός σύμβολος. Δηλαδή θα πρέπει, με συγχωρείτε, είναι κάπως δύσκολο να συνεχίσω γιατί υπάρχει θόρυβο στην αίθουσα. Ο πρόεδρος κάτι λέει στους ε, βουλευτές που συζητούν. Κύριε Φώση, κύριε Σβιεύκα, Παρακαλούμε, κάντε ησυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμπαθάτε με, συνάδελφοι, λέει η συγκεντρία. Και επίσης ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει είναι πώς ορίζεται το γενικό συμφέρον. Πώς θα χαρακτηριστεί κάποια πράξη που γίνεται για να προστατευτεί αυτό το συμφέρον. Τι πρωτοβουλίε καλύπτονται. Ιδιωτική πρωτοβουλία, ή όχι. Άλλο θέμα. Πώς γίνεται αυτή η καταγγελία. Εδώ σε, ε, στις εθνικές ρυθμίσεις έχουμε πολλές ε, ε, περιπτώσεις, ποιος κάνει την καταγγελία, ποιο την αποδέχεται, τι γίνεται στη συνέχεια και πώ μπορούμε ταυτόχρονα να έχουμε αυτή την καταγγελία σε αρμόδιες αρχές και να υπάρξει εγγύηση ανωνυμίας. Να μην υπάρχει υποχρέωση αποκάλυψης ταυτότητας του καταγγελόντος και όσον αφορά ε, επίση ε, το πώς θα επισημαίνεται κάτι γενικά στον κόσμο, στα μέσα ενημέρωσης, στο ευρύτερο δηλαδή κοινό, ε, έρευνα και έτσι να είναι δυνατόν να γνωστοποιείται σε όλες τις διαστάσεις μια φόρτη κατάσταση Μπορεί να έχουν περιπτώσει συκοφαντία βέβαια, ψευδείς καταγγελίες και αυτό να το ρυθμίσουμε και να υπάρχει επομένω μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή αρχή που να ασχολείται με όλα αυτά άλλο θέμα. Τι είδους προστασία, είπαμε προστασία της ανωνυμία, ε, αντίπεινα, πιέσεις, προστασία της θέση εργασία, προστασία της ε, αμοιβή και επίση τι θα γίνει όταν κάποιο σύρεται ενώπιον δικαστήριο και εκεί θα πρέπει να υπάρχει προστασία γιατί εναντίον του είναι κάποιε τεράστιε επιχειρήσει, έχουν τρομερού ε, νομικού συμβούλου. Οπότε κάποιον τρόπο έχουμε ε, δικονομική παρενόχληση ας πούμε. Οπότε θα πρέπει αυτόν τον καταγγέλλοντα να τον προστατεύσουμε γιατί κινδυνεύει, γιατί η, ε, η, είναι σε πολύ αδύνατη θέση τέλος πάντων. Και θα πρέπει Επίση να μπορεί να κρατήσει τη δουλειά του και ενώ γίνεται αυτή όλη η διαδικασία, ενώ βρίσκεται στο επίκεντρο του τυφώνα, θα πρέπει να μπορεί να επιζήσει. Ποτέ είναι και το θέμα της οικονομικής υποστήριξης, αλλά και το πώς θα πλαισιωθεί αυτή η κατάσταση, πριν έχουμε ε, καταχρηστικές ε, ρυθμίσεις. Άρα, οικονομική προστασία λέω εγώ, ώστε όσο η ζωή του είχε προστατευτεί να προστατεύεται ο καταγγέλων. Συμφωνήσαμε για τους βασικούς στόχους, βασικέ βασικές αρχές και είδαμε επίση ότι οι λεπτομέρειες ε, είναι αντικείμενο των ανταλλαγών απόψεων με τους συναδέλφους και θα δουλέψουμε και στο μέλλον μαζί. Ευχαριστώ. Thank you, and uh, thank uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, κυρία Ροζιέρ, για την εξαιρετική αυτή εισαγωγή. Και εγώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποιες ιδέες από την άποψη της Σουηδίας. Έχουμε ένα πολύ καλό και θεσμοθετημένο πλαίσιο για την προστασία των καταγγελτών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και βεβαίως χρειάζεται και θα είναι καλοδεχούμενη μια ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία θα συμπληρώσει αυτή. Βεβαίως έχει σαν σκοπό το ελάχιστο επίπεδο προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέποντας και αφήνοντας τα κράτη-μέλη αν θέλουν να είναι πιο φιλόδοξα και πιο αυστηρά όσον αφορά την προστασία αυτή. Πρόκειται για μια οριζόντια πρόταση οδηγίας που καλύπτει όλες τους τομείς της αγοράς εργασίας, τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε, η Επίτροπος Γιούραβα είπε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούλη στο Συμβούλιο για οριζόντια οδηγία. Πρέπει εμείς σαν Κοινοβούλιο όμως να το ζητήσουμε με επιμονή. Βεβαίως χρειάζεται προστασία κάθε είδους, ανωνυμία, έτσι ώστε να μην ε, είναι εξαιρετικά δύσκολο για ένα καταγγέλτη να αναφέρει διάφορες παραβιάσεις και όχι μόνο για παράνομες συμπεριφορές αλλά και άλλου είδους καταχρήσεις θα πρέπει να καταγγέλλονται. Πολλές φορές βλέπουμε σήμερα και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα να μην ε, υπάρχουν μόνο παράνομες δραστηριότητες. Πρέπει επίσης να προστατεύσουμε τους καταγγέλτες από αντίπεινα στο χώρο εργασίας, αλλά και γενικότερη προστασία ε, όταν αυτοί το χρειάζονται. Ο κύριος Καβαντά. Ευχαριστώ. Επιτέλους, το κείμενο αυτό που αφορά την προστασία ατόμων που βοηθούν το δημόσιο συμφέρον. Ήταν ε, πάρα πολύ χρήσιμη η δουλειά αυτή. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια, την κυρία Ροζιέρ, για πολύ επικοδομητική στάση που έχει κρατήσει. Δεν πρέπει να υπάρξει σε καμία περίπτωση σύγχυση μεταξύ ενός καταγγέλτη που προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και κάποιου ο οποίος ε, κάνει κάτι τελείως διαφορετικό, ο οποίος ε, ε, διαρρέει και διανέμει πληροφορίες για ιδιωτικό συμφέρον, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση ο ορισμός να είναι σαφής και να γίνει διαχωρισμός σαφής μεταξύ αυτών των ε, δύο κατηγοριών. Ο καταγγέλτης πρέπει να προστατεύεται από τη στιγμή που πλήττεται το δημόσιο συμφέρον, η δημοκρατία που καταγγέλει την διαφθορά. Η διαφθορά, όπως, ξέπετε, όπως ξέρετε, στην Ευρώπη είναι κάτι που πρέπει να καταπολεμήσουμε στην Ευρώπη. Χρειάζονται λοιπόν μέτρα για την προστασία αυτών των ατόμων από ανεξάρτητες δομές. Οι πληροφορίες θα πρέπει να επαληθεύονται με εμπιστευτικό τρόπο, να είναι ανώνυμες, να προστατεύονται δηλαδή τα άτομα αυτά που με θάρρος εκτίθενται εκθέτουν την οικογένειά τους, την θέση εργασίας τους και ξέρετε πολύ καλά ότι στην Ευρώπη δεν βρήκαμε τρόπο να προστατεύσουμε τον κύριο Σνόντεν, ο οποίος κατήγγειλε πρακτικές παράνομες της ε, Αμερικής δεν είμαστε σε θέση στην Ευρώπη, επαναλαμβάνω, να προστατεύσουμε τον κύριο Σνόντεν, ο οποίος αναγκάστηκε να καταφύγει σε μια πρεσβεία. Τώρα, θα πρέπει επίσης να μπορεί να προειδοποιείται ο παραβάτης πριν δημοσιευθούν τα στοιχεία που αφορούν ε, την εγκληματική του πράξη. Πρέπει επίσης να προστατεύσουμε τους καταγγέλτες από κάθε κίνδυνο. Δεν θέλω να επανέλθω. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να προστατευτεί η προσωπική του ζωή, η φήμη του, η εργασία του και η ατομική του ακαιρεότητα. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν και κάποια μέτρα προστασίας και κάποια οικονομική προστασία και ανταμοιβή. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να ε, δίνεται ένα αντίτιμο για αυτές τις πληροφορίες. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μεγάλη σημασία λοιπόν έχει και η προστασία του οικογενειακού και άμεσου περιβάλλοντος του καταγγέλτη Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι το θέμα αυτό ήρθε προ συζήτηση. Ελπίζω η Ευρώπη να μπορέσει να προστατεύσει αυτούς που εργάζονται για το κοινό συμφέρον και το κοινό καλό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αντικαθιστώ την σκιώδη συγγήτρια, την Κωνστόνς Λεγκρίπ. Γι' αυτό και θα πάρω το λόγο εξ ονόματός της. Η κυρία Λεγκρίπ θα ήθελε να σας υπενθυμίσει ότι με την οδηγία Trade Secrets ε, ήταν για πρώτη φορά ε, αναφέρθηκε ότι οι δραστηριότητες ε, τέτοιου είδους καταγγελιών παρέπει να προστατεύονται ε, τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εγκρίνουμε ένα οριζόντιο νομικό μέσο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα είναι η νομική βάση ενός τέτοιου νομικού ε, μέσου. Γι' αυτό το λόγο η κυρία Λεγκρίπ επικροτεί την πρόταση αυτή γιατί θεωρεί ότι αποτελεί μια προσπάθεια ορισμού ενός τέτοιου μέσου και, μέσου και αποφασιστικών ε, βημάτων για να βρεθεί η κατάλληλη νομική βάση αν υπάρχει βέβαια. Θα ήθελε η κυρία Λιγκρίπ να υπενθυμίσει σε όλο τον κόσμο ότι οι νομικές διατάξεις για τους καταγγέλλοντες, κάτι το οποίο είχε συζητηθεί και στην οδηγία, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει με τη δέουσα επιμέλεια για το κατά πόσο ε, θα πρέπει να ε, συμπεριλάβουμε ε, τρίτα μέρη και τα συμφέροντά τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πάρα πολλά έχουν υποθεί. Ε, συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν ε, και ήδη αυτό το θέμα ε, το είχαμε θέση ήδη ε, στην οδηγία που αφορούσε την εμπιστευτικότητα των ε, επιχειρήσεων. Ε, τότε το θέμα, από τότε το θέμα ήταν πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να επιμείνω επί ενός θέματος. Υπόθηκε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε πραγματικά ότι η προστασία των καταγγελόντων είναι ένας πυλώνας δημοκρατίας στον 21ο αιώνα. Γιατί, Γιατί από τη μία μπαίνουμε σε μια κοινωνία που είναι όλο και περισσότερο τεχνική και στο εσωτερικό των διαφόρων δομών μπορούμε να γνωρίζουμε ένα θέμα ε, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το γνωρίζουμε όταν είμαστε απ' έξω και το ξέρει πολύ καλά και ο Ζω Μαρί Καβαντά. Οι καταγγέλλοντες ε, είναι οι εγγυητές ε, της ελευθερίας του τύπου και της προστασίας των πηγών για τους δημοσιογράφους που είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Αν το δικαίωμα του τύπου το ε, ε, ε, δίκαιο του τύπου δεν προστατεύεται στην Ευρώπη, το δίκαιο της έρευνας είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύεται. Προστατεύουμε τους δημοσιογράφους που κάνουν έρευνες για πολύ σημαντικά θέματα. Ε, δεν θέλω να πω τίποτε καινούριο, έχουν τα περισσότερα υποθεί. Θα ήθελα να επιμείνω στο γεγονός ότι δεν πρόκειται να νομοθετήσουμε επί του κατά πόσο θα ανταμείψουμε ή όχι τους καταγγέλλοντες, αλλά να του τους προστατεύσουμε. Αυτό είναι το αντικείμενο της νομοθεσίας μας, να ε, πλαισιωθεί το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, όπως σε κάποιες επιχειρήσεις ε, προστατεύουμε τους συνδικαλιστές ή όσους υπερασπίζονται το συλλογικό συμφέρον, τουλάχιστον να μην διώκονται γι' αυτό. Πρέπει να ληφθεί υπόψη και το είπατε κι εσείς, ε, και αυτό είναι ο στόχος των καταγγελόντων, είναι η προάσπιση του συλλογικού, του γενικού συμφέροντος. Πρέπει να προστατεύσουμε εκείνον που διακινδυνεύοντας τη δουλειά του και ε, ποινική ε, δίωξη ε, προσπαθεί να προστατεύσει την δημοκρατία μας η οριζόντιος χαρακτήρας, η, βασική, η νομική βάση, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε ε, γιατί θα δημιουργούσε ε, πολλά ερωτηματικά αλλά εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στη Βυρζινή και στο σύνολο των σκιωδών εισηγητών για να προχωρήσει το κείμενο αυτό. Μία ακόμη φορά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και θα είναι ακόμη σημαντικότερο κατά τα επόμενα έτη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Μπορούμε... Α, κυρία Ρέντα, σας ξέχασα, συγγνώμη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπάρχει συνένεση και στην Επιτροπή μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα ότι υπάρχει ανάγκη οριζόντιας νομοθεσίας. Κάτι να σχολιάσω το οποίο ετέθη στη συζήγηση. Πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχει μία διαφοροποίηση νομικώς μεταξύ μίας καλοπροαίρετης και κακοπροαίρετης καταγγελίας το καρφί ας πούμε ε, που ακολουθεί ε, το δικό του ε, που προσπαθεί να προστατεύσει το δικό του συμφέρον και μόνο ε, είναι γεγονός ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι επιβλαβές για τους καταγγέλλοντες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τι γίνεται στο δικαστήριο, αν κάποιος πρέπει ενώπιον δικαστηρίου να εξηγήσει και να αποδείξει ότι είχε καλές προθέσεις ε, αποκάλυψης των πληροφοριών, με την αποκάλυψη των πληροφοριών αυτό συνήθω. Η άλλη πλευρά, ο εργοδότης, θα προσπαθήσει να ε, αποδείξει ότι είχαν άλλα κίνητρα ή άλλες άλλους στόχους ε, και ακόμη και για έναν καταγγέλλοντα που τελικά είχε ε, καλή πρόθεση, το να περάσει από αυτήν ε, την δικαστική διαδικασία είναι κάτι το οποίο καθένας θέλει να αποφύγει. Κανένας δεν θέλει κάποιος να αρχίσει να ερευνά τις προθέσεις του και να προσπαθεί να τις να τους, ε, να, να, να, δείξει, να τους δυσφημίσει ας πούμε ενώπιον του δικαστηρίου. Εγώ λοιπόν δεν καταλαβαίνω ποια είναι, ποιος είναι ο λόγος της διάκρισης. Ε, δημιουργεί μια ηθική ε, υποχρέωση που φαίνεται ότι είναι πιο σημαντική από το λόγο για τον οποίο μίλησε ένας καταγγέλων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να βασιζόμαστε στην πληροφορία που αποκαλύφθηκε και όχι στην πρόθεση του καταγγέλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, και εγώ ευχαριστώ. Ήταν η τελευταία ε, παρέμβαση για το θέμα αυτό. Θα ε, συνεχίσουμε με το σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, που είναι η ανταλλαγή απόψεων ε, για την απόσπαση εργαζομένων. Κυρία Γκούτελαντ, έχετε το λόγο. Thank you, Chair. This is the... Ευχαριστώ πολύ. Είναι η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων ε, για ε, την νομική ε, βάση για την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών αύριο ε, θα γίνει ψηφοφορία και θα ήθελα να ε, σας <coughs> καταθέσω κάποιες σκέψεις για αυτή την πάρα πολύ σημαντική γνωμοδότησή μας. Καταρχάς, πιστεύω ότι πρέπει να ε, προσέξουμε τους κύριους λόγους για τους οποίους γίνεται αναθεώρηση της, απόσπασης, της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων Θέλουμε να υπάρξει σωστή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης προώθησης ελευθερίας, παροχής υπηρεσιών και της ανάγκης προστασίας ε, των δικαιωμάτων των ε, αποσπασμένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καθορίσει αυτό το διτό στόχο στην πρότασή της. Υπάρχει μια σαφής ανάγκη επέκτασης ε, της προσπάθειας αυτής ε, αν η οδηγία ε, καταφέρει να πετύχει αυτή την ισορροπία. Η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λάβει μέτρα για να επιτύχει την κοινωνική βιωσιμότητα. Η διασυνοριακή, η ελεύθερη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και η κυκλοφορία των εργαζομένων, η απόσπαση αυτών δεν είναι ε, αντίθετα το ένα με το άλλο, αλλά συμμετέχουν στην ελεύθε, στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ε, αυτό προτείνουμε ε, την διαγραφή της νομικής βάσης, την οποία όχι να, όχι να την διαγράψουμε, αλλά να προσθέσουμε το άρθρο 153 α ε, και β και το άρθρο 153.2 δεν υπάρχει κανένα νομικό ε, πρόβλημα για τη συμπερίληψη αυτών των δύο ε, στοιχείων αν δεν συμπεριληφθούν ο διτός αυτός στόχος που ετέθη δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί στο μέλλον και δεν θα, θα δημιουργήσει προβλήματα στην ομολογία του δικαστηρίου. Ε, κάποιες επιχειρήσεις ε, δυστυχώς κάνουν κοινωνικό dumping για να μειώσουν το κόστος και να εκμεταλλεύσουν ε, να εκμεταλλευτούν τους εργαζομένους ως φθηνό εργατικό δυναμικό δημιουργώντας λοιπόν τη νέα νομική βάση 100, άρθρο 153 αβ και ε, το άρθρο 153.2 σημαίνει ότι ελαμβάνουμε πολιτική ε, ευθύνη όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων για την ίση αμοιβή για ίση εργασία, κάτι το οποίο χρειάζεται για να μην υπάρχει ε, διαφορετική χρήση ε, προδιαγραφών εργατικού δικαίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καβαντά. Όλοι γνωρίζουν ότι το θέμα αυτό είναι δύσκολο και η Επιτροπή μας θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ούτως ώστε το τελικό κείμενο το οποίο θα εγκριθεί να εφαρμοστεί και να έχουμε έτσι ουσιαστική πρόοδο και να φοβούνται λιγότερο από αυτό στις πατρίδες τους οι εργαζόμενοι και λέμε για δύο και σβάζει διαφορετικού είδους ονομοδιότητα εναρμόνιση από τη μια μεριά είναι το πώς δηλαδή τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να μεταφέρουν στην ένωμη τάξη αυτό το ευρωπαϊκό νομοθέτημα. Όπως πρέπει. Και αυτό θα πρέπει και εμείς να δούμε πώς θα ισχύσει και όσον αφορά τη συνθήκη για λειτουργία της Ένωσης προβλέπει ρητός ότι αν έχουμε διπλό στόχο για κάποια πρόταση θα πρέπει αυτό να γίνεται ε, ισορροπημένο. Και αν κάτι είναι κυρίως τώρα δευτερεύουν, τότε θα πρέπει να υπάρχει ενιαία, μία μόνο νομική βάση που να στηρίζει την πρόταση. Και να είναι βέβαια πρωταρχικό σκοπός. Τώρα, όσον αφορά την ε, νομική βάση για τους αποσπασμένους εργαζομένους, είναι η αρχή τη ελεύθερη κυκλοφοριασμένων, η ελευθερία της ε, εγκατάστασης και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Αυτό όμω δεν μα διευκολύνει και τόσο πολύ, ούτε αυτό το οποίο προσδοκάται τροποπληρώσει νομικής, νομική. Η κοινοτική αρμοδιότητα δεν είναι ίδια όταν έχουμε θέματα κοινωνική πολιτική και από την άλλη μετά θέματα ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή ελευθερία εγκατάσταση. Άλλη δυσκολία. Έχουμε το άρθρο 154 το οποίο πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπει να γίνει καμία διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Οπότε έχουμε το 153 ελληνική πολιτική για αυτό το λόγο. Οπότε εδώ προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει αυτή τη διαβούλευση. Και αν δεν ακολουθεί αυτή η διαδικασία, δεν μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση οπότε και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η επιλογή της προσθήκης της δεύτερης νομικής βάσης σημαίνει ότι αναπέμπεται η πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως πρέπει να το κάνουμε, αλλά έτσι δεν έχουμε ευελιξία. Δεύτερη νομική βάση σημαίνει «Α, να απόμπει προσωπικά». Δεν θα ήθελα να φρενάρουμε την πρόοδο της υπόθεσης αυτής. Γιατί και αυτό το θέμα την κοινή γνώμη σε όλα τα κρατημέλη και όλοι γνωρίζουμε ότι τώρα η Ευρώπη θα πρέπει να αποκτήσει πιο ξεκαθαρό κοινωνικό πρόσωπο, να είναι πιο ανθρώπινο. Άρα, να μην σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε αυτό το θέμα από τις δύο οπτικές γωνίες που είπαμε. Άρα χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, χρειάζεται περισσότερη ισότητα όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Άρα το κείμενο αυτό είναι εύστοχο από αυτή την άποψη. Και δεν είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει να έχουμε ως μόνο στόχο την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δεν νομίζω ότι αυτό θα αρέσει τόσο στους ε, Ευρωπαίους. Το αντίθετο. Οπότε θα πρέπει να τολμήσουμε να παρεκτείνουμε την νομική βάση. Εμείς θα πρέπει να προλιάνουμε το έδαφος ως οι ευρωβουλευτές. Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να αναζητήσουμε την ισορροπία στο κείμενο. Και έτσι, με ίση μεταχείριση, με ισόρροπο τρόπο, να έχουμε αυτές τις δύο νομικές βάσεις και έτσι να προχωρήσει το σχέδιο κοινών. Ε, εγώ νομίζω σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να κινηθούμε, κυρία εισηγητή. Ο πρώτος πρέπει να είστε σύντομοι διότι ήδη πήγε πέντε. Κύριε Φως. Ευχαριστώ. Το ΕΛΚ δεν πρόκειται να στηρίξει τη διεύρυνση εδώ αυτή τη νομική βάση. Και αυτό για πολλού λόγου. Πρώτον, ο στόχο αυτή τη πρόταση είναι να υπάρξει γενικότερη διεύρυνση, δηλαδή αποσπασμένοι εργαζόμενοι, είναι απλώς ένα μικρό κομμάτι της πρότασης. Ποιος είναι ο κεντρικός στόχος αυτού του κειμένου. Δεν αφορά τους αποσπασμένους ε, εργαζόμενους. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια οδηγία που αφορά την εσωτερική αγορά και η οποία πάβει να ισχύει. Βλέπουμε επίσης ότι το κράτος μέλος που επιθυμεί μπορεί να αυξήσει το επίπεδο προστασίας και το κράτος που θέλει να μειώσει το επίπεδο προστασίας μπορεί επίσης να το κάνει. Ε, αυτό είναι κάτι που το αφήνουμε στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών και η νομοθεσία των κρατών μελών που είναι αρμοδιότητα στους τομείς αυτούς των κρατών μελών θα παραμείνει. Είναι το θέμα της επικουρικότητας είναι καθαρά αρμοδιότητα των κρατών μελών αυτή που στοχεύει η οδηγία Είναι λοιπόν για μας λάθος αυτό που πάει να γίνει, γιατί κινδυνεύει να υπονομευθεί το όλο κείμενο. Ακριβώς αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Ο κίνδυνος λοιπόν της διεύρυνσης αυτής της νομικής βάσης είναι το όλο οικοδόμημα, το όλο νομοθετικό κείμενο να καταρρεύσει. Είναι ακριβώς αυτό που είπε και ο συνάδελφος Ζωμαρή Καναντά. Η διεύρυνση της νομικής ε, βάσης θα πρέπει να γίνει ξεκινώντας από μια νέα εξ ολοκλήρου νέα διαδικασία από το μηδέν, συμπεριλαμβάνοντας τους τομείς αυτούς που μας ενδιαφέρουν. Με αυτό τον τρόπο όμως όχι. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η τροποποίηση της οδηγίας που αφορά τους αποσπασμένους εργαζόμενους είναι πάρα πολύ σημαντικός όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τρόπος που θα επιλέξουμε να λύσουμε αυτό το θέμα θα αυξήσει ή όχι την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πάρα πολλές παρόμοιες περιπτώσεις όπου αγνοούμε τις κοινωνικές συνέπειες στην εσωτερική αγορά. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και πρέπει να δούμε αν πρέπει ή όχι να διευρύνουμε την νομική βάση όπως το προτείνει ο συγητής. Η ομάδα μας θα στηρίξει αυτή την πρόταση για διεύρυνση της νομικής βάσης όσον αφορά τα προς, την ε, προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Πρέπει να ξαναδούμε βεβαίως όλες τις λεπτομέρειες. Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο με αυτό το θέμα. Δεν λέω να το ξαναρχίσουμε από την αρχή, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να κοιτάξουμε τις αρνητικές συνέπειες και το θέμα των εργαζομένων που θέλουν να εργαστούν σε μια άλλη χώρα είναι καθοριστικό για την εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σάιερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αρχική έκθεση εμπεριέχει πολλά τμήματα που και στην Νομική Επιτροπή αλλά και σε άλλες επιτροπές προκάλεσε πάρα πολύ έντονη συζήτηση και εδώ και στα κράτη-μέλη. Η διεύρυνση της νομικής βάσης για αυτή την νομοθεσία θα διευρύνει ακόμα περισσότερο αυτές τις διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή θα εντείνουμε τις διαφορές, θα τις ενισχύσουμε και δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Η αρχική πρόθεση, όπως είπε και ο κύριος Βος, είναι να συμπεριληφθούν όλες αυτές οι προτάσεις στο κείμενο. Αυτή ήταν η αρχική πρόθεση για να ε, διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν προσθέσουμε και άλλα στοιχεία, 153 κτλ. Εδώ δημιουργούμε πολύ περισσότερες επιπλοκές. Το κείμενο γίνεται πολύ περίπλοκο. Είναι θέμα, αν θέλετε, που μας ε, υπέβαλε η Επιτροπή Απασχόλησης. Μας ζητάει αν ναι ή όχι μπορούμε να στηρίξουμε την διάβριση της νομικής βάσης. Εδώ υπάρχουν και κάποια κρυφά όμως αν θέλετε ερωτήματα. Εάν ναι ή όχι θέλουμε να προσθέσουμε νέα στοιχεία στην αρχική πρόταση, νομοθετική πρόταση της Επιτροπής που ξεπερνούν αυτήν την σημερινή νομική βάση. Τελικά βλέπουμε ότι τελικά αυτό που μας ρωτάνε είναι αν ναι ή όχι αρκεί αυτή η νομική βάση για την υπάρχουσα ε, νομοθετική πρόταση. Εμείς σαν ε, νομική επιτροπή είναι σαν να απαντούμε υποθετικές ερωτήσεις. Ερωτήσεις που δεν μας έχουν τεθεί ξεκάθαρα. Η ερώτηση για την νομική βάση θα πρέπει να μας τεθεί συγκεκριμένα και τότε θα απαντήσουμε. Αλλά υποθετικά και γενικά προτείνω να μην απαντήσουμε. Ας παραμείνουμε σοβαροί, ας διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας και ας μην προσπαθούμε να απαντήσουμε σε υποθετικές ή πλάγιες ερωτήσεις, οι οποίες δεν τίθενται ευθέως στην Επιτροπή μας. Αυτή τη στιγμή για το κείμενο που πρότεινε η Επιτροπή η νομική βάση αρκεί. Αυτό λέει η νομική μας υπηρεσία. Άρα, από νομική απόψεως και πολύ απλά, αν χρησιμοποιήσω το απλό επιχείρημα, η νομική επιτροπή δεν θα πρέπει να διευρύνει την απάντηση. Προς το παρόν, λοιπόν, ας αρκεστούμε σε αυτό, ας μην δημιουργήσουμε επιπλοκές οι οποίες ουσιαστικά θα φτάσουν στο αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που αρχικά ε, είχε η Επιτροπή Απασχόλησης. Βεβαίως ε, μπορούμε να συζητήσουμε και αυτό το θέμα, είναι πολύ ενδιαφέρον στη γενικότερη συζήτηση, αλλά σύμφωνα με το υπάρχον κείμενο δεν βλέπω για ποιο λόγο θα πρέπει να διευρυνθεί η νομική βάση. Εμείς σαν νομική υπηρεσία, ε, επιτροπή θα πρέπει να παραμείνουμε στη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας και να μην απαντούμε σε ερωτήσεις που δεν μας έχουν τεθεί άμεσα. Thank you. Ευχαριστώ. Όπως εξήγησε ήδη η κυρία Γκούτλαντ, θέλουμε διεύρυνση της νομικής βάσης για να καλύψουμε και τους δύο στόχους της προτάσεως και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών αλλά και το θέμα της κοινωνικής πολιτικής και όλα αυτά πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην νομική βάση. Άρχισε μια ματιά στην ε, γραμματοδότηση της νομικής υπηρεσίας, εξηγείται όπως εγώ το κατάλαβα, ότι έτσι είναι η ορθή μεθοδολογία. Και ορθό και δίκαιο. Άρα είμαι υπέρ της συζητήτριας. Καλώς λέει ο πρόεδρος. Δεν έχει ζητήσει άλλο τον λόγο. Και... Επομένως με αυτό το σημείο σαν ανταλλαγή απόψεων και σας ενημερώνω. Το σημείο υπαριθμών 10 αναβάλλεται. Για λόγους ελλείψης χρόνου. Αλλά αναβάλλεται και η ψηφοφορία για το 29 που είχε προβληθεί να γίνει και το αν δεν έχετε αντίρρηση Πάμε στο σημείο παριθμών 15. Πρόκειται. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ε, επειδή πρόκειται για περιορισμένη σύνθεση, πρόκειται για κεκλεισμένο θέλω συζήτηση, όποιος δεν δικαιούται να παραστεί,